Λοιπόν, εδώ προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τα μηχανήματα της ψηφοφορίας. Σε εξηγήσω το τι προσπαθούμε να κάνουμε. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Φαίνεται παράξενο σας λέω στα μέσα της εβδομάδας σας λέω καλή χρονιά, αλλά δεν έχω δει όλους σας. Και δεν είχα δει και όλους τους διερμηνείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά και από εμάς. Καλή χρονιά. Ελπίζω να είναι καλή χρονιά το 2018. Έχουμε μια μισή μέρα φορτωμένη. Έγκριση λοιπόν τη ημερήσια διάταξη. δεν έχω αλλαγέ να προτείνω. Έχετε εσεί, έχετε κάποιο πρόβλημα με την ημερήσια διάταξη. Όχι. Ευχαριστώ. Σημείο 2. Πρώτα απ' όλα, τεχνική φύσεως ζητήματα. Το πρόγραμμα για το 2018 για τι συναδριάσεις απεστάλλει ε, σε όλους σας και είναι και στην ιστοσελίδα. Ελπίζω να έχετε όλες τις ημερομηνίες της συνεδριάς επόμενης ε, να σημειώσετε τις ημερομηνίες. Την επόμενη Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου, στις 9 θα έχουμε κοινή συνεδρίαση της δικής μας Επιτροπής με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Εξωτερικών Υποθέσεων για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την, την συμφωνία την παγκόσμια για την νόμιμη μετανάστευση με την κυρία Κλάιν Σόλομον που είναι διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση. Αυτή είναι σημαντική συνεδρίαση την επόμενη πέμπτη το πρωί στις 9. Αυτά όσον αφορά τις τεχνικής φύσης ανακοινώσεις μου. Έχω μια θλιβερή και ταυτόχρονα χαρούμενη ανακοίνωση. Θλιβερή διότι όλοι θα γνωρίζετε ότι αυτή είναι η τελευταία συνεδρίαση της Άννα Κόφλιν που μετά από 16 χρόνια στην Επιτροπή ΔΕΒΕ πάει σε μια νέα θέση αναλαμβάνει τα καθήκοντά της την 1η Φεβρουαρίου Άρα είναι η τελευταία της συνεδρίαση. Δεν θα το γιορτάσουμε σήμερα. Τι 6.30 απόψε, σε αυτή την αίθουσα, μην το πείτε στις τεχνικές υπηρεσίες αυτό, έχουμε ένα ποτάκι. Για να ευχαριστήσουμε την Αν για τη δουλειά που έχει κάνει. 6.30 σε αυτή την αίθουσα, ε, μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών, θα είμαστε εδώ για να, σε αυτή την εκδήλωση να ευχαριστήσουμε την Άννα για τη δουλειά που έκανε εδώ επί σειρά ετών. Ήταν πολύ υπομονετική με όλους μας και ένα επικεφαλής μονάδας, Ντονατέλα Πρίμπα. Την ξέρετε πολλοί από εσά, γιατί έχει εργαστεί για, με θέματα ΑΚΕ και θα αναβάλει τα καθήκοντά τη την 5 Φεβρουαρίου. Δεν είναι εδώ, διότι έχει πάρει άδεια. Έχει κρατήσει άδεια την προηγούμενη θέση τη. Δεν είναι στην Επιτροπή μα θα την συναντήσουμε αρκετά σύντομα, σε περίπου δύο εβδομάδε. Εξήμιση απόψε, σημειώστε το παρακαλώ, η τελευταία σύνδεση επιτροπή Επιτροπής θα, θα πάρετε και σοκολατάκια. Λοιπόν, δεν το έχετε υπόψη. Λοιπόν, απόψε αυτό που σας είπα αργότερα. Λοιπόν, αυτό θα σας έλεγα, να χειροκροτήσουμε μάλλον. Αυτό σκεφτόμουν να καταγραφεί στα πρακτικά ότι ευχαριστούμε την ΑΝ για το έργο της επί σειρά ετών που μας βοήθησε με την εμπειρία στις, ε, να λάβουμε τις καλές αποφάσεις. Και αυτό να καταγραφεί στα πρακτικά παρακαλώ. <laughs> Δεν ξέρω να γράψεις εσύ αν τα πρακτικά. Α, ο γράφει τα πρακτικά. Λοιπόν, να καταγραφούν οι επίσημες ευχαριστήσεις Επιτροπής για το έργο της ΑΝ πίσω στη δουλειά μας. Σημείο 3, σημείο της διάταξης, τα πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων 9 και 10 Οκτωβρίου, 20-21 Νοεμβρίου και τα πρακτικά στο χαρτοφύλακά σας τα έχετε. Αν έχετε σχόλια, ενημερώστε τη γραμματεία σας παρακαλώ πριν τελειώσει η συνεδρίαση. Δεν έχουμε, αν δεν έχουμε παρατηρήσεις μέχρι τέλος θα θεωρηθούν τα πρακτικά κυκλήμα. Σημείο 4, ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχετε ανακοινώσεις, Ρωνο. Θα έρθει αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσοι ή άλλω. Οπότε μπορούν αύριο να το κάνουν. Και θα έρθει ο Γενικό Διευθυντή αύριο. Οπότε έχουμε διπλή δόση τη Γενική Διευθύνσεω Αρμοδία. Σημείο 5 απαλλαγή. Α, πάμε στι ψηφοφορίε. Συνήθω ξεκινάμε στι ψηφοφορίε τι Τετάρτε το πρωί στην Επιτροπή μα. Διαφορετική διαδικασία. Λοιπόν, απαλλαγή για το 2016. καταρχής ε, από πλευρά της ηγητού αν έχουν παρατηρήσεις για την γνωμοδότηση για την ε, απαλλαγή, τη θέση μας στην απαλλαγή, έχεις να πεις κάτι. Ρωτάω. Αν ο εισηγητής για την απαλλαγή θέλει να πει κάτι. Α, ψηφίσουμε λέει ο εισηγητής. Ωραία, ψηφίσουμε συνάδελφοι. Έχετε όλη την κάρτα σας. Θα κάνουμε πρώτα μια δοκιμή, να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Παρακαλώ πατήστε ένα κουμπί, να κάνουμε δοκιμή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εντάξει, δουλεύει το σύστημα, μπορούμε να ψηφίσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία 1. Α, υπάρχει πρόβλημα. Κάποια φορά έβαλα την κάρτα τη τράπεζα κατά λάθο και αναρωτιόμουν μέσα τι δουλεύει το μηχάνημα. Γίνονται αυτά. Λοιπόν. Λοιπόν, εάν θα είναι στην υπηρεσία για τις κάρτες για την ψηφοφορία, αν έχετε πρόβλημα με την κάρτα σας, το πείτε. Γιατί αυτό θα αναλάβει στη νέα τη θέση. Δουλεύει. Περιμένω να αλλάξει θέση ο κ. Νικολάζη που δεν δουλεύει το μηχάνημά του. Λοιπόν, λοιπόν η πρώτη ψηφοφορία, τροπολογία 1, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ παρακαλώ. Κατά,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 Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Τοπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία που άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Φουνσούλικα και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο σημείο 6, όπου ο κύριος Φουνσούλικα είναι και πάλι εισηγητής, απαλλαγή ο το 8ο, 9 10ο και 10ο ε, Ταμείο Ανά... Ανάπτυξη. Λοιπόν, ξεκινάμε τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την τροπολογία 4 παρακαλώ ξεκινάμε ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ κατά τα αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την τροπολογία 8 ξεκινάει η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για τη 14. Άρχεται η συμφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μικρή διαφορά. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για τη 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω ότι περνάει, αλλά θα δούμε. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά Να επαναλάβουμε. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας κάνουμε μια επαλήθευση για τη 17. Με μπερδεύουν σοσιαλιστές. Κουρνάνε τα χέρια τους πολύ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα το τροποποιημένο με νομιστική ψηφοφορία που ξεκινάει τώρα. Ψηφίσατε όλοι τέλος. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Συγητή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι τώρα. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους μάλλον. Σύντομος, λακωνικότατος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Σημείο 7, άλλη σημαντική έκθεση, ιδιαίτερα σημαντική, αφορά την προετοιμασία της θέση του Κοινοβουλίου για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Η είναι ο κύριο Ρούμπικ που είναι εδώ. Παουλ, θες να πεις κάτι πριν διεξαχθεί η ψηφοφορία. Yes, Και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τους καλούς συμβιβασμούς στους οποίους καταλήξαμε και στο συμβιβασμό 1 θυμάμαι ότι αντιστοιχεί με τη 14 αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σημαντική, όπως σας είπα, η ψηφοφορία αυτή. Ξεκινάμε την τροπολογία 1. Λόλα Σάντσες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές εξακρίβωση επαλήθευση για την 8 ξεκινάμε τώρα την ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας εντάξει ξε... απορρίπτεται λοιπόν τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ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 Έλεγχος για την συμβαστική 2α ξεκινάει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν. Τοπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τοπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τοπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την τροπολογία 27. Ξεκινάμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Λόγω ισοψηφίας. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για 35. Άρχεται τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 40 ξεκινάμε τώρα ψηφίσατε όλοι τέλος εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε τώρα στην τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 55 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες πέρας εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά έλεγχος για την 58 που ξεκινάει τώρα πέρας εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 η 60 καταπίπτει 61 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 61 νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε άρχεται ψηφίσατε όλοι απορρίπτεται λόγω ψηφίας. συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία ένα. λέει η πρόεδρος προφορική τροπολογία ένα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά έλεγχος των 72 έλεγχος των 72 λοιπόν ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 73 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 76 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές έλεγχος και για την 77 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 90 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται με μικρή διαφορά 91 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 91 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 96 άρχεται η ψηφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 103 άρχεται η ψηφορία 103 Ψήφισαν άπατες, πέρας. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχο για την 108 άρχεται η ψηφοφορία, νομίζω ότι απορρίπτεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 110 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε άπαντες, πέρας, εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 111 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 112 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Πέρας. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος για την 117. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές Έλεγχο για την 118, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 119. Ας ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. πέρα. Εγκρίνεται. Α, έχουμε και την προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον Παουλ Ρούμπικ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντική ψηφοφορία. Θα δούμε τι θα γίνει με τους συναδέλφους στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ, όσοι θέλουν να φύγουν, ε, παρακαλώ να αποχωρήσουν. Γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική νέα έκθεση που θα μας απασχολήσει με το πριν για ένα σημαντικό θέμα. Ένα θέμα που πριν από μερικά χρόνια όλοι θεωρούσαν ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών, να έχει επιληθεί θεωρούσαν όλοι, αλλά υπάρχουν τώρα νέα προβλήματα και χαίρομαι που θα συζητήσουμε το 8 η ενίσχυση της βιωσιμότητας ε, του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών. Πολύ σημαντικό θέμα. Η μας είναι ο κύριος Σαλ ε, Γκερένς. Σας παρακαλώ, όσοι αποχωρούν μπορούν παρακαλώ να συζητήσουν έξω από την αίθουσα. Έχει πολύ χώρο, έχει καφενεία. Παρακαλώ, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αν θέλετε να συζητήσετε, σας παρακαλώ ε, να επιτρέψετε στον εισηγητή μας να παρουσιάσει την έκθεσή του. Σάρλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας υποβάλλω την τελική μου έκθεση, τον τελικό μου σχέδιο έκθεσης και βεβαίως ε, θα ψηφίσουμε επ' αυτής. Ελπίζω να ψηφιστεί από την Ολομέλεια πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η έκθεση αυτή θέτει μια σειρά από θέματα. Ήδη τα εξηγήσατε κατά την προηγούμενη συζήτηση, δηλαδή κατά την εισαγωγή που κάνατε. Τονίσατε ότι η δανειοληψία και το χρέος είναι σημαντικό μέσο χρηματοδότησης των οικονομιών. Πολλές ε, αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα είχαν χωρίς αυτή τη δυνατότητα καμία δυνατότητα να επενδύσουν στην περαιτέρω και βιώσιμη ανάπτυξή τους. Στα πλαίσια του δημοσίου δανείου. Έχουμε από τη μία τους πιστωτές, τον πληθυσμό της χώρας ε, που λαμβάνει το δάνειο, τις τράπεζες, ε, τους καταθέτες, ε, τα κράτη που λαμβάνουν το δάνειο και τα δικά μας κράτη. Για παράδειγμα, αν μια δική μας τράπεζα με ασυνείδητο τρόπο δανείσει στο Νιζέρ, το κράτος μας υφίσταται τις αρνητικές επιπτώσεις. Και αν υπάρχουν πολλά τέτοια δάνεια, μπορεί να προκύψει μια τραπεζική κρίση, όπως ε, προέκυψε την περίοδο 2007-2008, ε, της οποίας κρίσης, τις επιπτώσεις, τις αισθανόμεθα ακόμη. Η υπερχρέωση αποκαλύπτει πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εάν ασυνείδητα ή ελαφρά την καρδία γίνονται αυτά τα δάνεια, οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο ότι χάνει ο δανειοδότης, Πολλές φορές τις επιπτώσεις την υφίστανται και οι κάτοικοι των χωρών που λαμβάνουν τα δάνεια. Υπάρχουν για παράδειγμα ε, τα προγράμματα θεσμικών προσαρμογών. Η συμφωνία της Washington που είχαμε την δεκαετία του 90 Έχουμε επίση τα δικαιώματα των καταθετών αλλά και τις υποχρεώσει. Και τα κράτη και οι τράπεζες όλοι έχουν και δικαιώματα και υποχρεώσει. Προσπάθησα λοιπόν να θέσω μερικέ βασικές αρχές που θα πρέπει να μας οδηγούν. Μπορεί να φαίνεται λίγο θεωρητικό αλλά δεν έχω στόχο να αποστασιοποιηθώ από την κατάσταση. Απλώ θέλω να πω ότι σε επίπεδο αρχών είναι αρκετά απλή η κατάσταση. Θεωρώ και νομίζω ότι είναι θεμελιώδης ε, αξία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι το δικαίωμα ε, ανάπτυξης είναι ανθρώπινο δικαίωμα όλων των πληθυσμών. Ναι μεν δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα πρώτης γενιάς, αυτά που προέκυψαν από την ε, Γαλλική Επανάσταση, αλλά παρόλα αυτά είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Μπορεί να μην έχουν ενταχθεί σε κάποιες διεθνείς συνθήκες, αλλά είναι βασικό θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Εάν λοιπόν, λοιπόν προκύψουν αντιθέσεις, όπου από τη μία έχει δικαιώματα ο δανειοδότης και από την άλλη η ικανοποίηση των δικαιωμάτων του θα σήμαινε ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο πληθυσμός της χώρας που έλαβε το δάνειο, Εάν απειλείται η ίδια επιβίωση αυτού του πληθυσμού, τότε νομίζω ότι το ανθρώπινο δικαίωμα ανάπτυξη πρέπει να υπερισχύσει των δικαιωμάτων των δανειοδοτών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα ο δανειοδότης. Έχει δικαιώματα, αλλά πρέπει να πλαισιωθούν καλύτερα αυτά τα δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν στο μέλλον να θεωρείται ότι κάποιες τράπεζες ε, είναι υπερβολικά σημαντικές για να χρεοκοπήσουν. Too big to fail. Πρέπει να ελέγξουμε εάν δανειοδότησαν ασυνείδητα. Πρέπει ε, να καταλάβουμε ότι αυτό έχει επιπτώσει στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, άρα και στον πληθυσμό των χωρών μα και στην κοινωνική του κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει πλέον να δίδονται δάνεια, αλλά πρέπει τα δάνεια να χορηγούνται με καλύτερο, πιο σωστό τρόπο το μόνο δάνειο που θα πρέπει να δίδεται είναι αυτό που θα εξυπηρετεί την ε, ανάπτυξη του πληθυσμού των χωρών που λαμβάνουν το δάνειο. Όταν πρόκειται για δάνεια που λαμβάνουν δημόσιες αρχές. Αυτές είναι οι βασικές αρχές επί των οποίων θέλω να τεθεί η έκθεσή μου. Η πιο συνηθισμένη κατάσταση αντιθέσεων είναι αυτή την οποία μόλις ε, περιέγραψα. Πρέπει λοιπόν το δικαίωμα στην ανάπτυξη να υπερισχύει του δικαιώματος ε, αποπληρωμής του δανείου. Και εάν υπάρχουν ε, απρόβλεπτες καταστάσεις που δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί από τις αρχές της χώρας ε, που έλαβε το δάνειο, τότε θα έπρεπε να υπάρχει μια διακοπή στην αποπληρωμή του χρέους αν υπάρξει θεομηνία, τσουνάμι, σεισμός κτλ. Επίσης, η πολιτική δανειοδότηση πρέπει να εγγράφεται στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης. Και γι' αυτό αναφέρω τα θεμελιώδη δικαιώματα του κράτους δικαίου, τις βασικές δημοκρατικές αρχές, οι οποίες στις χώρες μας ε, τουλάχιστον και νομίζω και σε αναπτυσσόμενες χώρες πολύ εμπνέονται από τα πρότυπά μας, θα πρέπει να είναι στο κέντρο των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου το δικαίωμα να συζητάει και να ψηφίζει τον προπολογισμό του κράτους τους. Αυτό είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Αλλά σε ορισμένα κράτη υπάρχει τόση διαφθορά και οι ηγέτες βλέπουμε ότι τα δάνεια που παίρνουν τα τρώνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής. Και αν το δικαίωμα αποπληρωμής τελικά υπερισχύσει, τις συνέπειες τις υφίσταται ο πληθυσμός. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπερισχύει το δικαίωμα στην ανάπτυξη, να υπερισχύει του δικαιώματος αποπληρωμής του χρέους. Γιατί αυτό θα παίξει αποτρεπτικό ρόλο και προς τους δανειοδότες. Δεν θέλουμε να δυσχεράνουμε την επιβίωση των δανειοδοτών, αλλά θα πρέπει να δρούν υπεύθυνα και να υφίστανται τις επιπτώσεις των ενεργειών τους. Και αυτό θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα πολυμερές πλαίσιο. Υπάρχουν ε, διάφορες αρχές που αντιμετωπίζουν τις κρίσεις της υπερχρέωσης. Για παράδειγμα, έχουμε το, τη Λέσχη των Παρισίων. Τα μέλη ε, της Λέσχης είναι τα κράτη είναι τα κράτη που έχουν λάβει και τα κράτη που έχουν ε, ε, δώσει δάνεια. Ε, η συμφωνία του Λονδίνου αφορά κυρίως τις ιδιωτικές τράπεζες, τις εμπορικές τράπεζες. Θα πρέπει λοιπόν κάπως να συνδυάσουν τις ενέργειές τους. Επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό και εξηγώ γιατί στην ανάλυση μου εξηγώ ποια είναι η θέση των κρατών μελών της Ένωσης γιατί δεν συμφωνούν πάντα. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν επικυρώσει ένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και γι' αυτό τονίζω ότι πρέπει να εγκρίνουμε τις αρχές της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την υπεύθυνη πολιτική στη δανειοδότηση και την ανάπτυξη, ούτω ώστε να υπάρχει κοινή ευθύνη και των δανειοδοτών και των δανειοληπτών. Αυτές είναι οι αρχές Τη ε, συνδιάσκεψη των Εθνών για την υπεύθυνη δανειοδότηση. Αλλά δεν έχει επικυρώσει αυτό το ψήφισμα και καταγγέλουμε την ε, άρνηση του Συμβουλίου μέσω της κοινή του θέσης για την αναδιάθρωση του δημοσίου χρέους που είναι κρίθη, όπως είπα από την πλειοψηφία στα Ηνωμένα Έθνη. Η θέση της Ευρώπης μπορώ να πω ότι βασίζεται σε μη ομολογούμενες ε, επιδιώξεις των κρατών μελών. Θα πρέπει να υπερβούμε αυτήν την προσέγγιση. θεωρώ ότι οι αρχές ε, της ανάπτυξης πρέπει να είναι η βάση της πρόθεσής μας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση, ούτως ώστε αυτές οι αρχές να γίνουν δεσμεύσεις. Έχετε λοιπόν ένα σύνολο από άρθρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα για να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις ε, στάσεις πληρωμών των κρατών μελών. Αντίστοιχες διατάξεις ε, για τις πτωχεύσεις, τις εμπορικές πτωχεύσεις υπάρχουν στα εθνικά μας δίκαια. Θα έπρεπε να υπάρχει κάτι παρόμοιο σε επίπεδο ένωσης και κρατών μελών. Θέλω βέβαια να ακούσω και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει μια λευκή βίβλο, να κάνει μια, έναν απολογισμό της κατάστασης και να κάνει προτάσεις για το μέλλον. Καταλήγοντας. Δεν θέλω να παρανοηθώ. Λέγοντας ότι δεν πρέπει να δίδονται ανεύθυνα δάνεια. Δεν εννοώ ότι θα πρέπει να σταματήσει η δανειοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών. Έχουμε δέσμευση ως κράτη-μέλη και ως Κομισιόν να πάει στο 0,7 του ΑΕΠ μας ε, η δημόσια βοήθεια προς την ανάπτυξη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με δάνεια. Θα πρέπει να γίνει και με ε, χορήγηση ε, πιστώσεων. Γι' αυτό λέγεται δημόσια βοήθεια προς την ανάπτυξη. Δεν θέλω λοιπόν πολλά κράτη-μέλη να μην μπορούν πλέον να λαμβάνουν δάνεια. εάν δεν δοθεί κάποιο δάνειο. Δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ανάπτυξη μιας χώρας. Και αν μια χώρα δεν μπορεί πλέον να λάβει δάνεια, θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει βοήθεια. Με βάση τα κριτήρια του ΩΣΑ. Αλλά εάν κάποια δάνεια απλώς ε, πλούτησαν τους διεθαρμένους δικτάτορες, δεν είναι δυνατόν ε, μετά να ισχυρίζονται ότι βοήθησαν την ανάπτυξη της χώρας τους. Όλα αυτά προφανώς δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Ορίστε οι προτάσεις μου, είναι πολύ σύντομες, βασίζονται στην προσπάθεια επίτευξης αποτελεσμάτων. Ξέρω και πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε περαιτέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε, να εστιάσουμε σε αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα ανάπτυξης των πληθυσμών και αυτό να υπερισχύει της αποπληρωμής του χρέους. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του παρελθόντος, κάτι που εξακολουθεί να είναι λεπτό θέμα και να δημιουργήσουμε και τις βάσεις για μια πολιτική μέλλοντος, για να αποφευχθεί η επανάληψη των κρίσεων που είχαμε στο παρελθόν. Επανειλημμένα το συζητήσαμε όταν εξετάσαμε την κατάσταση των τριών χωρών που επλήγησαν από τον ιό έμπολα, τότε είχαμε διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε επαρκής ανάπτυξης του σχολικού τομέα, ε, της υγείας, της διοικητικής ικανότητας του κράτους για να μπορεί να εκτελεί τις λειτουργίες του ως κράτος. Όλα αυτά κατά πολύ ενίσχυσαν την κρίση. Άλλες χώρες γειτονικές όπου δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, δεν υπήρχε αυτή η έλλειψη χρηματοδότηση τη ανάπτυξη, όπω στη Σενεγάλη για παράδειγμα, στην Ιγυρία, υπήρξαν ε, κάποιες, ε, κάποια κρούσματα, αλλά πολύ σύντομα αντιμετωπίστηκαν. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θεωρώ ότι και η Κομισιόν πρέπει να λάβει πρωτοβουλίε και να επιτύχει να πει στα κράτη-μέλη να σημειωθεί πρόοδο επί του θέματο αυτού και σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σοβαρό το θέμα και έχουμε τώρα μια σειρά από σκοδησικητές και πρώτος ο κύριος Σένφιλ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θέλετε το λόγο? Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. No tak jak Pani Przewodnicząca zapowiadając ten temat powiedziała. Και... Όπως ε, είπατε στην αρχή, το θέμα αυτό είναι δυσχερές και επίμαχο. Και νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από αυτού. Ακόμη και ο εισηγητής ε, παρουσίασε τις διαφορετικές απόψεις επαυτού. αυτού. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι απόλυτα ανοιχτός. Το περιεχόμενο της έκθεσης δεν μας δημιουργεί προβλήματα γενικά. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους συνεργάτες του που μας υπέβαλαν αυτό το κείμενο. Είναι πολύ ισορροπημένο, έλαβε υπόψη όλες τις απόψεις και τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από πλευράς και του δανειοδότη και του δανειολήπτη. Και το βασικό θέμα που τονίζει ο συγητής είναι οι κοινωνίες των χωρών. Το πρόβλημα, ξέρετε, είναι, είναι ότι υπάρχουν δύο μέρη. Από τη μία μεριά οι πιο ισχυροί, αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, είναι οι δανειοδότες που έχουν τα κεφάλαια και δίνουν δάνεια. Και από την άλλη μεριά είναι οι αρχές των χωρών που λαμβάνουν τα δάνεια που αποφασίζουν πόσα θα αξιοποιήσουν, για ποιο λόγο και τι ύψος ε, δάνειο θα ζητήσουν. Όλα αυτά ε, βασίζονται στην αρχή της ανάπτυξης των χωρών, αλλά όπως ανέφερε και ο συγητής, πολύ συχνά τα δάνεια αυτά μπαίνουν στις τσέπες ε, κάποιων. Για παράδειγμα, ηγετών αυταρχικών κρατών και ο πληθυσμός παίρνει μόνο ψίχουλα. Τα δάνεια λοιπόν δεν εξυπηρετούν τους στόχους που θα βοηθούσαν την ανάπτυξη των χωρών. Πολύ σωστό το παράδειγμα της επιδημίας έμπολα. Αν δεν υπήρχε η βοήθεια από πλευράς της Ευρώπης αλλά και άλλων των ΗΠΑ κτλ τότε, τότε το ερώτημα αν θα είχε επιζήσει κανείς στις χώρες αυτές γιατί την επιδημία αυτή τη σταμάτησαν οι δυτικέ χώρες και όχι οι υγειονομικές αρχές των χωρών αυτών που σχεδόν δεν υφίστανται. Τώρα, για την έκθεση. Υπάρχουν κάποια θέματα που θεωρώ ότι είναι επίμαχα και ο Σέλκ θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα συμπεριφερθούμε Να πω λοιπόν τα θέματα που μας δημιουργούν προβλήματα και μετά θα σας πω με ποια συμφωνώ. Τώρα, το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ομοσπονδική Γερμανία δεν ε, στήριξαν το ψήφισμα αυτό. ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Κάποιους λόγους έχουν. 41 χώρες συνολικά απέσχον. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Πρέπει τόσο πολύ να τονίσουμε το θέμα αυτό, αυτού του ψηφίσματος. Δεύτερον, αναφέρεστε σε διεθνείς μηχανισμούς για να αντιμετωπιστεί το θέμα της υπερχρέωσης. Κοιτάξτε, το η σύστημα χρηματοδότησης των κρατών ε, του αναπτυσσόμενου κόσμου είναι περίπλοκο, δεν ε, προκύπτει από μία πηγή. Διάφοροι όμιλοι μπορεί να χρηματοδοτούν τις χώρες αυτές, ε, διάφοροι, διάφορες κοινοπραξίες δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και τις περισσότερες φορές οι δανειοδότες είναι ιδιωτικέ εταιρείε που έχουν μετόχους. οι οποίοι επενδύουν, ξέρετε, το κεφάλαιό τους για να ε, κερδίσουν κάτι. Τώρα λοιπόν κάποιος θα τους αποφασίσει, θα αποφασίσει για αυτούς τι θα γίνει με τις επενδύσεις τους, με ποιους όρους θα δανειοδοτούν, με ποιους όρους θα λειτουργούν αυτοί οι ιδιωτικοί φορείς. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Και επίσης, αυτή η ιδέα του κοινωνικού ελέγχου σε αναπτυγμένες κοινωνίες όπως οι δικές μας οι δυτικές χώρες αλλά ακόμη και σε αναπτυσσόμενες θα έπρεπε πάντα η βάση να είναι ο κοινωνικός έλεγχος. Είμαι πεπισμένος όμως ότι οι πολίτες των χωρών αυτών οι περισσότεροι τουλάχιστον ε, δεν μαθαίνουν τι δάνεια λαμβάνουν οι χώρες τους και πώς χρησιμοποιούνται και δεν γνωρίζουν ε, τους όρους αποπληρωμής του δανείου. Πώς θα καθορίσουν τους όρους αυτούς. Να καθορίζει η κοινωνία κάποιους όρους που μετά θα είναι υποχρεωτικοί. Βεβαίως, Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση το, του πληθυσμού για τους στόχους των δανείων, για τους όρους και τις προθεσμίες αποπληρωμής. Αυτό θα έπρεπε να είναι προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου. Ναι, αλλά αυτό ξέρετε δημιουργεί προβλήματα. Κυρίως ε, θα έπρεπε να παίζουν ρόλο τα κοινοβούλια. Δεν θα αποφασίζουν βέβαια για τα πάντα τα κοινοβούλια, γιατί οι κυβερνήσεις κυρίως αποφασίζουν για την ε, λήψη δανείων και φέρουν και την πολιτική και ποινική ευθύνη. Αλλά αν υπήρχε κάποια πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούσε να ενημερωθεί η κοινή γνώμη δηλαδή τι ύψους είναι τα δάνεια που έχουν ληφθεί από μια χώρα και ποιες είναι οι περίοδοι αποπληρωμής τους, αυτό θα ήταν χρήσιμο. Και κάτι ακόμη. Ο εισηγητής έθεσε επανειλημμένα την αρχή ότι το ανθρώπινο δικαίωμα της ε, ανάπτυξης των κοινωνιών θα πρέπει να υπερισχύει των αρχών της ε, αποπληρωμής των δανείων, της αρχής της αποπληρωμής των δανείων. Ως γενική ιδέα είναι θαυμάσια, πολύ ανθρωπιστική, αλλά νομίζω ότι τελικά είναι αιμονική γιατί ξέρετε οι αρχές αποφασίζουν και όχι οι πολίτες, οι αρχές κυρίως των κρατών αυτών που στις περισσότερες περιπτώσεις τη χώρες αυτές είναι αυταρχικές, ορισμένες φορές και δικτατορίες. Αυτοί παίρνουν τα δάνεια και μετά τα στέλνουν στο λογαριασμό τους στην Ελβετία ή σε κάποιο νησί και μετά λένε μετά θέλετε να πούμε ότι ωραία να ε, ακυρώσουμε τα δάνεια αυτά. Οπότε τα χρήματα αυτά των διαφόρων σατραπών αυτών μένουν στους λογαριασμούς τους, ε, στους παραδείσους φορολογικούς και τα παιδιά του κόσμου ε, παραμένουν φτωχά ενώ τα δικά τους πηγαίνουν στα καλύτερα πανεπιστήμια. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν για τις επιπτώσεις ε, αυτών που προτείνουμε. Μπορεί να ακούγονται πολύ όμορφα, πολύ ανθρωπιστικά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ντόρο Φουντζούλιβε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα πρώτα. Συγχαρητήρια για το σχέδιο της έκθεσης προς τον κύριο Γκέρνς. Και βλέπουμε στην ιδεολογική έκθεση ότι το θέμα ε, δεν είναι αργιστή το χρέος, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες δεσμευτικοί για την υπόθεση αυτή και έτσι να επιληθεί αυτό το πρόβλημα του υπερβολικού χρέους και να μην υπάρχουν ε, εκτροπές. Οπότε τώρα έχουμε τα κατάλληλα μέσα, τις κατάλληλες διατάξεις που όμως δεν έχουν αρκέσει ούτως ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση του χρέους και ιδίως ε, να υπάρξουν συνθήκες που να ευνοούν την ανάπτυξη. Ε, γι' αυτό λοιπόν και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το ότι εδώ ε, αναδεικνύεται ένας μόνιμος μηχανισμός διαχείρισης του χρέου των χωρών και να υπάρχει και ένα πολυμερές νομικό πλαίσιο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια αναδιάρθρωση αυτού του δημόσιου κρατικού τέλο πάντων χρέου. Οπότε σα τονίζω ότι για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του χρέου θα πρέπει να έχουμε διαπραγματεύσει για την που θα πρέπει να γίνουν αμελητή και αποτελεσματικά και επίση να καταλήξουν σε κάποιο είδου σταθεροποίηση ε, του χρέους και το παράλληλα να προστατεύσουμε την βιώσιμη οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη επίσης και τώρα κάτι άλλο το οποίο θέλω να σας προτείνω είναι σε σχέση με την βιωσιμότητα του χρέους. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στις σκέψεις του οικονομικού άξονα. Θα πρέπει να δούμε επίσης ε, τι άλλε επιπτώσει υπάρχουν από το βάρος του χρέους, τη δυνατότητα τη χώρα να μπορεί να τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια που έχουμε σημαντική αύξηση του χρέου και στον ιδιωτικό τομέα και στο κράτος στι αναπτυσσόμενε χώρες. Θα πρέπει να προβληματιστούμε περαιτέρω όσον αφορά το πώς μπορούμε να καλύψουμε τις επενδύσεις σε κάποιο είδους ε, τομείς κλειδί όπως παιδεία, υγεία, οικονομία και υποδομές. Και επίσης σας υπενθυμίζω ότι το δάνειο είναι σημαντικό μέσο ούτω ώστε να στηρίξει επενδύσεις. Άρα η βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και η σχετική στόχη είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή να κάτσουμε να κάνουμε κάποιο αξιολόγηση του τι γίνεται με αυτό το χρέος για τις υπερχρεωμένε χώρες ακριβώ να λάβουν υπόψη αυτούς τους στόχους και έτσι να δούμε προτεραιότητα ε, πώς θα έχουν τα δικαιώματα του δανειστού, τέλος πάντων δανειοδότη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε την Τζούντι τη Αρχεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκίνησα μαζί με το θέμα λέγοντας ότι ε, θεωρήσατε ότι έχει περάσει αυτό το θέμα και εγώ έτσι θυμάμαι ότι είχε γίνει μια μεγάλη εκστατεία για την ε, πέτειο του ορόσημου του 2000 σε σχέση με το υπαχθές χρέος κλπ. Και θυμάμαι το 2005 την Glen Eagles τότε που όλοι προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε το χρέος. Οπότε και είπαμε ότι όλα αυτά είναι πια περασμένα, είναι στο χρονοτούλαπο. Ε, τώρα πρέπει να το ξανοίξουμε το χρονοτούλαπο γιατί είμαστε ενώπιον μιας νέας κρίσης χρέους. Άρα τη σωστή ώρα ήρθε η έκθεση του κύριου Γκέρνς και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι ελκύει πάλι την προσοχή μας το ζήτημα αυτό. Οι, οι πράσινοι θα κατεβάσουν κάποιες τροπολογίες πρώτα-πρώτα για την ε, διαφάνεια. Ξέρουμε ποιος, τι και σε ποιον δανείζει και με βάση ποια κριτήρια. Είναι υγιές, είναι λογικό υπό τέτοιε συνθήκε να δανείζει κανεί από τι χώρε άλλο θέμα που έχει σχέση όμως τι γίνεται με τα εμπορεύματα και τους ε, φυσικούς πόρους, πρώτες ύλες γιατί μίλησαμε για το ότι παίρνουν μεγάλα δάνεια αυτές οι χώρες επί τη βάση αυτών των ε, πόρων που έχουν αλλά που ακόμα δεν έχουν εξοριχθεί ούτως είναι ακόμα στο έδαφος και οι τιμές φουσκώνουν ας πούμε τι γίνεται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο ή τι γίνεται με το πετρέλαιο στο τσάδ τότε που τελικά οι τιμές καταποντίστηκαν. Όμως κατεβλήθη το δάνειο και θα πρέπει να αποπληρωθεί σε είδος. Άρα τα ξέρουμε που γίνονται τα λάθη και θα πρέπει να λαμβάνονται. Άλλο. Blending. Ανακάτεμα. Με βοήθεια με δανειοληπτική ικανότητα. Μα αυτό οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερο δανεισμό. Τι κίνδυνοι ελοχεύουν, τα λέμε και τα ξαναλέμε πολύ καιρό αυτά. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς οι πράσινοι συμφωνήσαμε για αυτό το Ταμείο Εξωτερικών Επενδύσεων που είναι κάτι το θετικό και προσπαθήσαμε αυτό να το πλαισιώσουμε με ένα σωρό ρήτρες ούτως υπήν εξασφάλισης, αλλά να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος του να βυθιστεί στο χρέος και πάλι μία αναπτυσσόμενη χώρα. Θα πρέπει να δούμε πριν από τις τροπολογίες ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος των εξορυκτικών βιομηχανιών όσον αφορά το χρέος. ή ITS, δεν λέμε τώρα μην σας ζελίζουμε τα αρχικά. Οπότε τελικά αυτό γίνεται ένα εργαλείο, ένα μέσο για τους ε, δανειστές. Όμως δεν μας βοηθάει ούτως ώστε να έχουμε διαφάνεια που να διακρίνει τα συγκεκριμένα δανεία. Τέλος πάντων, μπράβο στον κύριο ε, Γκέρενς και θα συμβάλλουμε και εμείς. Λόλα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα συγχαρητήρια προς τον κύριο Γκέρενς γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογο το σχέδιο κειμένου. Συμφωνούμε με τις βασικές γραμμές του και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναδεικνύει το κείμενο ότι δηλαδή το δικαίωμα της ανάπτυξης θα πρέπει να κατησχύει του δικαιώματος του δανειστού. Άρα δεν θα πρέπει αυτό το χρέος να είναι μέσω υπόταξης αυτού του των, των χωρών, των πιο φτωχών. Ε, γι' αυτό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο προτύπων ούτω ώστε να υπάρξει ένας ορισμός του τι είναι υπεύθυνο δάνειο με κριτήρια ανεξάρτητα, δίκαια και επίσης έτσι να κρίνεται το θεμητόν, το νόμιμο και το βιώσιμο του χρέους αλλά πρέπει να δούμε επίση ποιε είναι οι ανάγκε των ε, προσώπων, των, του, κόσμου και τι γίνεται με τα επαχθή χρέη. Επίση να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη στον αυτοκρατικό χρέο. Ε, άρα χρειάζεται διεθνή μηχανισμό και έτσι να υπάρξει κάποια ανάλυση που να εστιάζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα κατεβάσουμε τροπολογίε. θα συμβάλλουμε στο κείμενο, να κάνουμε κάποιες ε, ε, διευκρινήσει που υπάρξει διαφάνεια, πάρα πολύ βασικό, τόσο ώστε να υπάρχουν σωστά δάνεια. Επίσης θα πρέπει να τηρηθούν στα πλαίσια του σημείου του g και της Αντισαμπέμπα οι υποχρεώσεις να τηρηθούν όσον αφορά το βιώσιμο χρέος. Και επίσης θα πρέπει να δούμε το πώς τα δάνεια για το τα συγγνώμη, οι πληροφορίε, τα δεδομένα για το δάνειο πρέπει να πάρουν σε κάποιο μητρό προσβάσιμο. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα δάνεια των εξωμένων χωρών, γιατί είναι σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε εκθέσει για όλα τα δάνεια, ιδιωτικά και δημόσια προ τι αναπτυσσόμενε χώρε. Και επίση, θα πρέπει να δούμε όσον αφορά τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τι γίνεται. Πώς γίνεται αυτό το blending, αυτή η ανάμειξη. Τι γίνεται με αυτά τα νομικά πρόσωπα. Γιατί θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ρήτρες εξασφάλισης όσον αφορά τις αρχές και να μην έχουμε υπονόμευση της ο πληρωμής του χρέους. Πολλές φορές κάποιες επενδύσεις είναι καμουφλαρισμένα δάνεια, οπότε τις σωρεύεται. Τα έχει πει αυτό ο ΣΕ. Γιατί συνήθως λέει ο ΣΑ ότι το 84% του χρέους δεν επιδέχεται αποπληρωμή. Είναι αδύνατο να αποπληρωθεί. Είπαμε είναι θετικό το κείμενο του εισηγητή και θέλουμε τελικά να καταλήξουμε σε κάποια πολυαξιόλογη έκθεση της Επιτροπή μας. Λόλα, ευχαριστούμε και εγώ θέλω να λάβω το λόγο και να σας πω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα που είπε η Λόλα για το ότι θα πρέπει να πριτανεύσει διαφάνεια σε σχέση με την εκταμείευση αυτών των ε, δανείων. Δεν πρέπει τελικά να ωφελούνται οι διεφθαρμένοι. Αλλά έχουν ευθύνη και οι τράπεζε. Αφού δανείζει τον κόσμο, θα πρέπει να έχει κάποια ιδέα για το πώ θα πληρωθεί το χρόνο. Δεν δανείζει επί τη βάση του πιανού. Μα, πληρώνουμε τώρα και ανεβαίνει η τιμή του εμπορεύματος λες. Μα τελικά όμως πέφτει η τιμή. Μην δανείζονται δισεκατομμύρια επί τη βάση του ότι θα ανέβει η τιμή του εμπρόσωπου, όπως η κυρία Σαρχεντίνη. να κανεί δεν έχει στοιχεία ότι είναι δυνατή η αποπληρωμή. Α, πάω στην τράπεζα να ζητήσω ένα στεγαστικό δάνειο, κάτι να φτιάξω στο σπίτι, ναι, αλλά η τράπεζα τι θα πει. Θα πει, το κάνεις αυτό, θα πει η τράπεζα, και έχει προσθέμενη αξία για το σπίτι σου. Α, και στην Μοζαμβίκη δύο τράπεζες. Δάνεισαν στην κυβέρνηση να φτιάξει αλληλευτικό στόλο. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Πήγαν σε περάκτης offshore. Τα κτήματα κανένας δεν ξέρει που πήγαν. Οπότε έχουμε τώρα διάφορα θεσμικά όργανα διεθνή τα οποία δεν δένουν στην μοζανδική Ε, και γι' αυτό έχει πληγεί πάρα πολύ το μέρο των δημοσίων υπηρεσιών. Έχει δίκιο ο κύριο Γκέρνς. Ήρθε η ώρα να πούμε, α μην ξανά έχουμε μια κρίση σαν το Ιωβρίο του 2000. Μα το 2005 είχα την Κίνοκ που ε, προείδρευε σε εκείνη την ισομερή συνέλευση για τη ΣΑΚΕ και είχαμε αυτή την ολομέλεια και βλέπαμε τις διαφάνειες και αυτό μου φαίνεται σαν χθε. Ε, ας μην ξαναζήσουμε τα ίδια. Για να δούμε. Τι θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα πει η υπηρεσία εξωτερική δράση. Για να το κοιτάξουν το Πάλι τώρα για το blending. Δεν ξέρω. Έχουμε βγάλει τίποτα συμπεράσματα. Έχουν πάρει κανένα μάθημα. Γιατί και στη δική μου χώρα ο ιδιωτικό τομέα έχει εμπλακεί πάρα πολύ. Όχι μόνο σε μεγάλα έργα, αλλά κάνουν και υπεργολαβία βασικές υπηρεσίες. Και είδατε τι έγινε με την κατάρρευση των εταιριών που είχαν πολύ σημαντικές ε, συμβάσεις. Πού πήγαν αυτές οι υπηρεσίες. Οπότε τώρα η κυβέρνηση στον τομέα της υγείας είναι αντιμέτωπη σημαντικά προβλήματα. Τα νοσοκομεία δεν καθαρίζονται. Όλοι αυτοί που το ανέλαβαν για το τίμημα που πήραν δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Τρομερές οι συμβάσεις που εκχωρήθηκαν. Οπότε τι κάνουν, συμπιέζουν τις τιμές, δεν μπορούν τους εργαζομένους, συνθήκες τραγικές και τελικά δεν μπορούν να εκπληρώσουν τη σύμβαση. Ε, ε να καταλάβουμε. Τι έγινε με την Καρίλιον, στον Ιωμένο Βασίλειο, τι έγινε στη Μοζαμβίκη. Να, τι είπα να πει το blending και η υπεργολαβία των κρατικών υπηρεσιών γιατί ακούμε για χρηματοδότηση, για το blending, αλλά μάθαμε τίποτα από όσα γίνανε. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Να βλέπω και για μια πρωτοβουλία τώρα η Credit Suisse έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτά γιατί είχαν ανακατευτεί αυτά στην υπόθεση εκείνη της και λένε τώρα για κάποιο σύμφωνο διαφάνειας α, τα είπε πάρα πολύ καλά η Λόρα ας υπάρξει επιτέλους κάποιο μητρό, κάποιο πρωτόκολλο για αυτά τα δάνεια δανείζουν για κάποιο έργο το οποίο ποτέ δεν υλοποιείται πολύ σοβαρά θέματα κάτι πρέπει να κάνουμε δεν ξέρω έχει κάτι υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει Ποιο άλλοι ζήτησαν το λόγο. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Από την Ντεύκο. Πρώτα πρώτα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σαν Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ θεωρούμε πρόσδεκτη αυτή την έκθεση και τη διεξαγωγή της συζητήσεως επί του θέματος. σημαίνουμε αύξηση του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών και φτάνουν σε επίπεδα χρέους που πλησιάζουν αυτά που είχαμε όταν έπρεπε να αναλάβουμε διάφορες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έχουμε ανησυχητικέ τάσεις, εξηγούνται σε κάποιες περιπτώσεις. Πήγα στη Μοζαμβίκη ήδη εδώ και κάποιους μήνες. Πήγα για να αναλύσω ποιες είναι οι συνέπειες καταστάσεως της Μοζαμβίκης, που επικρατεί στη Μοζαμβίκη στην απτυξιακή πολιτική μας, διότι επηρεάζεται η πολιτική μας. Τονίζει τις ανησυχητικέ τάσεις η έκθεση και είναι σημεία από συζήτηση ενδιαφέρουσα. για βιώσιμη ανάπτυξη χρειάζεται η χρέωση, αλλά πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Να υπάρχει το σωστό πλαίσιο δανειοδοτήσεων. Οτι ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη και υπεύθυνη δανειοδότηση και δανειοληψία. Συμφωνούμε λοιπόν με την έκθεση ότι η δυνατότητα διαχειρίσεως του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών χρήζει ενισχύσεως. Πρέπει να καταγράφονται στοιχεία. Χρειάζεται να συντάσσονται εκθέσεις, να γίνεται ανάλυση των στοιχείων. Χρειάζεται σωστή στατική διαχείριση του χρέους, να επικρατεί η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική η διαφάνεια. Εκεί επικεντρώνουν προσπάθεια. Η δανειοδότηση και η δανειοληψία χρειάζεται πλαισίωση. Χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία το θέμα. Πρέπει να βασιστούμε επί των ισχυουσών αρχών των G20. Αρχές που εξέφρασαν οι G20 το 2017 και τις UNCTAD επίση το έργο χρησιμοποιεί βάση. Χρειάζεται σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών αυτών οι επενδύσεις, οι κρατικές προμήθειες είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και χρειάζεται και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και χρηματοοικονομική πολιτική και ξανά, επαναλαμβάνω, η διαφάνεια σημαντική. Η συζήτηση να βάνει χώρα επίσης και στην προσπάθεια για την βελτίωση ε, των εσωτερικών οικονομικών και της δυνατότητα εισπράξεων αυτών των χωρών ε, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και εντάσσεται στο γενικότερο θεματολόγιο το φορολογικό. Παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το χρέος των αντισωμένων χωρών. Είναι βασική μας εντολή αυτή. Έχουμε δραστηριοποιηθεί. Χρησιμοποιούμε διάφορες προσεγγίσεις. Συνεργαζόμαστε με την Παγκόσμια Τράπεζα και με το μέσο αυτής για τη διαχείριση του χρέους. Μέσο που στηρίζουμε. Έτσι βελτιώνεται η δυνατότητα της διοίκησης να χειρίζεται το χρέος της. Η κυβέρνηση διαχειρίζεται καλύτερα το χρέος της. Το χρέο δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, είναι αναγκαίο, χρειάζεται όμω η ορθή διαχείριση αυτού. Και να χρησιμοποιείται για του σωστού σκοπού εθνική πολιτική. Θέλουμε να συνάβουμε και στην ανάλυση τη UNCTAD και το σχετικό σύστημα τη UNCTAD για διαχείριση του χρέου. Επιτρέψει αναπτυσσόμενε χώρε και στι χώρε εν γέννη αυτό το σύστημα να διαχειρίζονται το χρέο του. Να βελτιώνουν τι δυνατότητε πρόβλεψη ε, της βιωσιμότητας του χρέους τους. Σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζουμε υποστήριξη των προπολογισμών. Θα συζητήσουμε ξανά στη Γενική Διεύθυνση το θέμα αυτό. Μακροοικονομική σταθερότητα είναι μία από τι βασικέ αρχέ της πολιτικής για υποστήριξη του προϋπολογισμού. Θέλουμε να παρακολουθούμε και τι γίνεται στις χώρες από πλευράς μακροοικονομικής πολιτικής. Συνεργαζόμαστε με το Δούνο του για χώρες. Θέλουμε να, μέσω της υποστήριξης του προπολογισμού να έχουμε καλύτερο έλεγχο. Να βελτιωθεί και έλεγχος των εθνικών κοινοβουλίων. Σε όλες τις συζητήσεις τονίζεται και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων. Αυξάνουμε τις προσπάθειες για την κινητοποίηση εσωτερικών μέσων για πράξεις και έσοδα των χωρών. Συνεργαζόμαστε και με τον ΟΣΑ για τη διαφάνεια στο Παγκόσμιο Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών. Συνεργαζόμαστε το θέμα του blending και πώς αυτό συνδέεται με τα εξωτερικά επενδυτικά προγράμματα είναι σημαντικό. Συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους συναδέλφους μας. Ούτως ώστε η βιωσιμότητα του χρέους αντιμετωπίζεται σωστά να γίνονται σωστέ σωστές επενδύσεις. Θέλουμε να δούμε τι είδους δανειοδότηση θέλουμε να υφίσταται και ποιο επίπεδο δανειοληψίας. Συνεργαζόμαστε στενά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα για τη βιωσιμότητα του χρέους. Εν γέννη, ευπρόσδεκτη συζήτηση που θα διεξαχθεί επ' αυτού, τροφή προσκέψη και προσβελτίωση των συστημάτων δεν λέω ότι τα πάντα είναι τέλεια, πόρο απέχει η κατάσταση από αυτή. Υπάρχουν καταστάσεις άκρως ανησυχητικέ. Είμαστε όμως έτοιμοι να συνεργαστούμε το Κοινοβούλιο επί της εκθέσεως και να προβληματιστούμε περαιτέρω πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Χουσέιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προφανώς υποστηρίζουμε και εμείς την έκθεση και την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πολιτική σκοπιά. Αναφερόμαστε στη στρατηγική για την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λέμε ότι θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω δημόσια χρηματοδοτήσεως. Χρειαζόμαστε και άλλες προσεγγίσεις, χρειαζόμαστε δάνεια και χρέη για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους στόχους της ε, παγκόσμιας αναπτύξης και άλλες πηγές χρηματοδοτήσεως που θα χρηματοδοτούν τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως είναι το εμπόριο, ε, ξένοι άμεση, ε, άμεσες επενδύσεις κατά πολέμηση των παρανόμων ροών χρημάτων. Υποστηρίζουμε λοιπόν το θεματολόγιο της Αντίσαμπέμπα όσον αφορά την εξασφάλιση περισσότερων πηγών χρηματοδιώτησης για την επίτευξη των στόχων βιωσίμου αναπτύξεως. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και η δανειοδότηση όπως αναφέρεται όμως στην έκθεση και όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δανειοδότηση αυτή πρέπει να είναι υπεύθυνη και όχι ανεύθυνη, η ΔΕΜΗ αν, ε, ε, εάν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης θα αποτύχουμε. Υποστηρίζουμε την έκθεση λοιπόν. Υποστηρίζουμε και τις πρωτοβουλίες που περιέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενθαρρύνουν μεγαλύτερη υπεύθυνη δανειοδότηση και προσβλέπουμε στις συνεχιζόμενες συζητήσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ να απαντήσω, να θέσω μια ερώτηση μα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει Πρόεδρος. Αναφερθήκατε στη Μοζαμβίκη και εξετάζει το θέμα στήριξη του προπολογισμού. Τι έγινε τελικά. Εγώ τι συναισθάνομαι. Αυτό που έλεγα. Ανεύθυνη κυβέρνηση παίρνει χρήματα από μια ανεύθυνη τράπεζα. Χωρίς να ελέγχει δίνει τα χρήματα η τράπεζα και τότε ο μόνο μου είναι να κόψουμε τη στήριξη του υπολογισμού που αφιερώνεται στι δημόσιε υπηρεσίε, Δεν πρέπει να εξετάσουμε στο μοντέλο μα, πώ θα κινηθούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Καταλαβαίνετε που το πάω. Αν περικόψουμε τη στήριξη του προπολογισμού, βλάπτεται η υγεία, οι δημόσιε υπηρεσίε κλπ. Η παιδεία. Ναι, περίπλοκο το θέμα, λέει η Κομισιόν. Αφορά εγγύσει που δίνονται για τα δάνεια και όχι τα δάνεια άμεσα. Οι εγγύσει που έχουν παρασκευθεί από την κυβέρνηση. Δεν έχει λήξει ιστορία. Ε, εκκρεμεί ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βοηθήσουμε τις χώρες άμεσα μέσω έργων και προγραμμάτων. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το τι θα κάνουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Στην περίπτωση της Μοζαμβίκης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τις ζητήσεις. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες αυτού και τι έχει κάνει η κυβέρνηση κλπ. Αλλά ζητήθηκε από την κυβέρνηση της Μοζαμβίκης να αναλυθεί δράση για περισσότερη διαφάνεια, να ερευνηθεί το τι συνέβη και να γίνουν τα δέοντα. Γνωρίζω που η για την Πρωτοβουλία περί διαφανείας, η ιδέα των τραπεζών, να υπάρχει ένα διεθνές σύστημα που θα ασχοληθεί με το θέμα. Στηρίζεται ένα τέτοιο σύστημα. Ξέρω ότι λέτε, έχουμε τη συζητήσει των G20, πολύ συχνά το κουβεντιάζουν και δεν γίνεται τίποτα. Ε, το θέμα είναι αν υπάρχει πραγματικό πνεύμα να προωθεί το θέμα. Απάντηση. Ήδη ε, γίνονται συζητήσει και με την Παγκόσμια Τράπεζα θα συμμετάσχουμε τον Μάιο στι Βρυξέλλε σε μια διάσκεψη. Η ιδέα τη υπεύθυνη δαδιοδότηση είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, είναι επίκαιρο και είναι κατάλληλη στιγμή. Και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη αυτή η έκθεση, διότι είναι πολύ καλή αυτή τη στιγμή για να συζητήσουμε τι ιδέες. Ευχαριστώ. Ενθαρρυντικό αυτό. Ίσως μπορούμε να μάθουμε περισσότερα αυτή η διάσκεψη για την υπεύθυνη αντιδότηση και να γνωρίζουν οι και να συμμετάσχουν εκεί. Ο κ. Γκέραν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που παρενέβησαν του ΕΛΚ, των Σοσιαλιστών, της ΓΚΟΕ, των Πρασίνων που υποστήριξαν που εξετίμησαν την έκθεση. Πόρο απέχει από το να είναι τέλεια αυτή η έκθεση, όμως έχει μόνη φιλοδοξία κάπως να μετακινήσει τις γραμμές και τα όρια. Συμμερίζεται ευρέω την ανάλυση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι ερμηνεύουμε παρομοίως τα πράγματα και τα φαινόμενα που εκτιλήσονται και που ίσως να αποκτήσουμε μεγαλύτερο εύρο στο μέλλον. Ας συνοηθούμε επί βασικών αξώνων. Λοιπόν, ερώτηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το άρθρο 14 του ψηφίσματος. Τι άποψη έχει από αυτού. Αναφέρομαι εκεί σε ένα ψήφισμα που υιοθετήθηκε με πλειοψηφία από τον ΙΕ. Ψήφισμα 10 Σεπτεμβρίου του 2015 ούτω ώστε να δημιουργηθεί μηχανισμός μόνιμος που θα χειρίζεται τις κρίσεις των αναπτυσσομένων χωρών. Αυτό το ψήφισμα προβλέπει μια εντολή που δεν έχει ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των κρατών μελών της θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την εντολή. Θα μπορούσαμε ήδη να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία ενεργοποίησης της εντολής, ώστε εν συνεχεία να μπορεί να δημιουργηθεί ένα νομικό πολυμερές πλαίσιο για την αδιάθρωση του κρατικού χρέους. Σε επίπεδο της παγκοσμίου διακυβερνήσεως, στον τομέα αυτό, έχουμε ένα ευχολόγιο μεγάλο που περιέχει τα πάντα. Πρέπει να γίνει κάποιος συντονισμός. Προσπάθησα να συμπεριλάβω τις δυνατότητες που υπάρχουν, που έχουμε ως κράτη-μέλη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ε, μετακινηθούν κάποιες οι θέσεις, προσπαθώντας να θέσουμε και όρια των δράσεων. Εξηγούμε. Η ανάπτυξη δεν είμαστε εμείς που θα οδηγήσουμε του τους λαούς αντισωμένων χωρών στην ανάπτυξη. Αυτοί θα πρέπει να αναπτυχθούν από μόνοι τους, Συζητώντα με τις κυβερνήσεις τους. Αυτό που μπορούμε να απαιτήσουμε και το κάνω στην έκθεση, στο σχέδιο εκθέσεω, είναι το εξή. Τα κοινοβούλια, τα κράτη-μέλη και τα, οι αναπτυσσόμενε χώρε, οι δανειοληπτικέ χώρε που κάνουν θα πρέπει να, ε, να ελέγχουν τα, ε, οι βουλές, τα κοινοβούλια αυτών των χωρών τα δάνεια που λαμβάνουν. Ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις αρχές τις δημοκρατικές μας και συνεργασίες. Θα πρέπει να τα πετούμε αυτά σε συνεργασία με αυτές τις χώρες. Εναλλακτικό τι θα είναι, να φλουμε έναντι μιας πρακτικής όπου τα χρήματα κυκλοφορούν και μπαίνουν στις τσέπες των διεφθαρμένων δίκτυων δικτατόρων και των φαρχικών κυβερνήσεων και θα πρέπει να πληρώσουμε μετά από 20 χρόνια πληθυσμοί τα χρήματα αυτά που δεν, οδη... δεν χρησιμοποιήθηκαν για τριξιακούς σκοπούς. και, λοιπόν, όταν δεν μπορούν να αποπληρωθούν τα χρέη. Λοιπόν, τα ποσά αυτά των... Ε, στα λογιστικά υπολογίζονται για τις χώρες αυτές ενώ δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Αυτό είναι κάτι ε, που δεν πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αφήσουμε πίσω μας οριστικά αυτή την πρακτική, αυτή την ιστορία. Σαφώς. Οι πιστωτές ε, που έχουν δικαιώματα. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Αυτοί οι πιστωτέ που δυνατηρούν ελαφρά την καρδία αυτέ τι χώρε όπου τα εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν λόγο, η θέση αυτών πιστωτών δεν θα πρέπει να ενισχύεται. Αντιθέτω, θα πρέπει να αποδυναμωθεί. Και γι' αυτό το λόγο η εφαρμογή, η δημιουργία συστήματος πολυμερούς που θα διαχειρίζεται τις κρίσεις των αναπτυσσομένων χωρών, τις κρίσεις χρέους των αναπτυσσομένων χωρών, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να το αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν, επειδή έχει αποτελματωθεί η κατάσταση, θα πρέπει να προωθήσουμε το ώστε να υπάρχει μία απεμπλοκή. Εδώ θέλουμε, δεν θέλουμε ε, θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε αλλιώς την ανάπτυξη, όχι να αποκλείσουμε κάποιες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προστασεύσει τις επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί μπορεί να, αυτό να έχει μορφή προγράμματος σχεδίου που τελεί υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διαφόρων φορέων αναπτύξεως εάν ε, δεν πληρούνται οι όροι τόσο ώστε η ίδια η χώρα μόνη της να τα εφαρμόσει θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι εναλλακτικέ λύσεις χρηματοδότησης. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις εναλλακτικέ λύσεις πριν αποκλειστεί κάποια χώρα. Και πρέπει αυτή να είναι μια αρχή δράσης μόνιμη. Ο Μαλρό είπε ότι εάν είναι, αφορείται μόνο το κράτος, αποκλειστικά το κράτος, είναι η αρχή του πολιταρχικού κράτους. Χρειάζεται ελάχιστο διακυβέρνησης το λένε στους G7, στους G20, στον ΟΣΑ. Χρειάζεται όμως να υπάρχει κάποια αρχή και τελικά σε τι χρησιμεύει ο Αυτοί για την ώρα βλέπω έχουν συντάξει τα πιο ευφυή κείμενα επί των οποίων μπορούμε να βασίσουμε μια παγκόσμια διαχείριση σε αυτό το, σε αυτό το τομέα. Όταν λοιπόν, όταν έκανε συγκεκριμένε προτάσεις ότι δεν θα πρέπει η ισχύ των πιστωτών ενισχύεται σε περίπτωση δανείων που χορηγούνται ανεξέλεγκτα και αναφέρομαι στο βελγικό δίκαιο. Δεν προστατεύει πλέον αυτούς τους πιστωτές το βελγικό δίκαιο. Ε, όπως ένα hedge fund που αγόρασε κάποιες πιστώσεις από την Αργεντινή στην τιμή 25-30% ονομαστικής αξίας. Αγόρασαν αυτές τις πιστώσεις για το 1 τρίτο της ονομαστικής αξίας. Μετά πήγαν στη Νέα Υόρκη και κατήγγειλαν την κυβέρνηση Αργεντινής υποχρώνοντας να ξεπληρώσουν πλήρως το δάνειο 100%. Και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Το βελγικό δίκαιο σε περίπτωση που θα μπορούσε να γενικευτεί σε επίπεδο 28 ήδη θα μπλοκάριζε. Μάλλον θα δημιουργούσε μια δύναμη που θα μπλοκάριζε αυτή την πρακτική Αυτά είναι κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε στο μέλλον περαιτέρω. Θα ήθελα ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Περισσία Εξωτερική Δράση να αναλάβουν την υποχρέωση να προτείνουν κάτι πιο στεναρό, ένα είδο λευκή βίβλου, πείτε το όπω θέλετε, ανακοίνωση, που θα, θα στριμώχνει τα κράτη-μέλη Υπάρχουν και τα κράτη-μέλη που θέλουν να κινηθούν και έχουν λάβει υποδειγματικά μέτρα. Θα πρέπει όμω να είναι υποδειγματική όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά για να συμμορφωθούμε με αυτά που αναφέρουμε στα κηρύγματά μας για το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, το σεβασμό του δημοκρατικού κράτους, το διαχωρισμό των εξουσιών κλπ. Τη διάκριση των εξουσιών. Αυτές είναι οι προτάσεις που έχω και χαίρομαι που οι περισσότεροι συνάδελφοι, σχεδόν όλοι, είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν την προσέγγιση μου. Περιμένω ανυπόμονα τις τροπολογίες σας. Κυρία Πρόεδρε, θα, θα σας πει το χρονοδιάγραμμα των επομένων σταδίων που θα ακολουθηθούν από την έκθεση. Ευχαριστώ απείρως, πολύ θερμά. Και προσβλέπω σε συζητήσεις που μας οδηγήσουν σε μια ολοκλήρωση της συζήτησης και να προωθήσουμε κάπως τις θέσεις μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, υπάρχει κάποια καθυστέρηση, ξέρω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Τέθηκε συγκεκριμένη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροπολογία, συγγνώμη, την παράγραφο 14. Και για το αν μπορεί να κάνει περισσότερη επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα αναφέρει στους ανώτερους το θέμα αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση καταψήφισε αυτό το ψήφισμα των ΗΠΑ. Μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ αυτό το θέμα, γιατί κατόπιν έχουμε μια κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, η Κομισιόν. Εργαζόμαστε μαζί με την Γενική Διεύθυνση για το θέμα αυτό που ασχολείται με την μακροοικονομική επιτήρηση. Επ' αυτού. Μας είπαν ότι όταν έγινε η συζήτηση το 2015 δεν θεώρησαν ότι ήταν ε, τα Ηνωμένα Έθνη το κατάλληλο πλαίσιο για να συζητηθεί το θέμα αυτό σε παγκόσμια βάση. Αυτή είναι η απόφαση που λήφθηκε τότε και εξακολουθεί να ισχύει. Αλλά ε, ακούσαμε τι είπατε και με χαρά να συνεχίσουμε τη συζήτηση και σημειώσαμε ότι θέλετε μία ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Θα ε, το αναφέρω αυτό στις άλλες υπηρεσίες και θα δούμε τι θα υπάρξει ως συνέχεια. Σαν πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Ξέρω την εξήγηση που είχε δώσει η κυρία Λούκας εκείνη την περίοδο εκ μέρους της Ένωσης. Ακόμη και αν εξακολουθεί να θεωρεί ότι ισχύει αυτή η εξήγηση, θεωρώ εγώ ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα μπορούσαν να είναι ο χώρος όπου θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι κατά τη συμβολής της Παγκόσμιας Τράπεζας, ε, του Δελτανή Ταφ και τα λοιπά. Και για το πιο φόρουμ είναι πιο κατάλληλο, ε, νομίζω ότι το Ηνωμένα Έθνη είναι το πιο κατάλληλο φόρουμ. Γιατί ε, είναι μέλη της σχεδόν όλες τις χώρες, έχει συγκεκριμένους ειδικευμένου οργανισμούς, ε, την ΚΝΟΥΣΕΝΤ, από εκεί θα μπορούσε να ξεκινήσει η πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί ένα πολυμερές νομικό πλαίσιο. Δεν ξέρω τώρα ποιο θα το ε, έχει ως αρμοδιότητα με τα Ηνωμένα Έθνη ή καποιο άλλος φορέας, αλλά κάπου πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση. Έτσι πρέπει να δουν το θέμα τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να υπάρξουν πολλές ασάφειες στην Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη όταν ε, ετίθεται το θέμα του να σεβαστούν τις δεσμεύσει του δεν λένε τίποτα. Σε όλε τι γλώσσε δεν λένε τίποτα. Πρέπει λοιπόν να το καταγγείλουμε αυτό ω Επιτροπή. Πρέπει να καταστεί σαφέ ποιο θέλει να σεβαστεί τι δεσμεύσει του. Να λοιπόν, μια νέα δοκιμασία στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν είμαι υπέρ τη υπερβολική ε, επιφυλακτικότητα τη Κομισιόν. Πρώτα να δει τι λένε όλοι και μετά να με σποβάλει πρόταση. Θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα πολιτικό τα κράτη-μέλη δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους, ορισμένα ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους συμφέροντα. Η πολιτική ανάπτυξη λαμβάνει όμως υπόψη και τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών. Συμφωνούμε με την προσέγγιση της Κομισιόν, αλλά θα ήθελα να αντιδράσουν με κάπως πιο αποφασιστικό τρόπο. Με συγχωρείτε που είμαι τόσο ειλικρινής. Και αν μπορείτε να παρακαλέσετε τους ε, προϊσταμένους σας, τους ανώτερούς σας να έρθουν εδώ, θα τους θα πω επίσης τα ράτα. Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, επιχειρήσουμε να συμβαδίσουμε. Ευχαριστώ Σάρλ, νομίζω ότι κατάλαβαν τι θέλεις να τους πεις. Προθεσμία για τροπολογίες 30 Ιανουαρίου 12. 13 μάλλον Φεβρουαρίου εννοούσε η πρόεδρος και θα ψηφίσουμε τέλος Φεβρουαρίου. Σημείο 9. Συγγνώμη, 30 Ιανουαρίου. Λοιπόν, έχουμε την έκθεση τώρα για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των εξωτερικών μέσων ε, χρηματοδότησης της Ένωσης. Εγώ είμαι η συντάκτρια της γνωμοδότησης για το θέμα αυτό είναι πολύ σύντομη. Υπενθυμίζω, συνάδελφοι, η ΑΦΕΤ κάνει μια έκθεση για τα δικά της μέσα. Εμείς, με εισηγητή τον κύριο Γερέρο, κάνουμε μια έκθεση για τα δικά μας μέσα. Δεν θέλω λοιπόν να μιλήσω για τα δικά μας μέσα στην γνωμοδότηση προς την ΑΦΕΤ και πώς θα πρέπει να δράσουν στο μέλλον. Αυτό θα μας το εξηγήσει ο Ενρίκε με την έκθεση που θα μας υποβάλει τον επόμενο μήνα νομίζω. Οι τροπολογίες λοιπόν, α μάλλον ε, δεν τροπολογώ την έκθεση της ΑΦΕΤ γιατί μόλις αυτή τη βδομάδα την είδα αναφέρει μερικά ενδιαφέροντα σημεία ζήτησα την, στην από την εισηγήτρια να έρθει σήμερα εδώ το πρωί αλλά δεν μπορούσε αναφέρει μερικά λοιπόν ενδιαφέροντα σημεία αλλά επειδή δεν ήθελα να κάνουμε διπλή δουλειά περιορίστηκα σε ορισμένες τεχνικές πλευρές της έκθεσης της ΑΦΕΤ για τους κοινούς εφαρμοστικούς κανόνες του κανονισμού που καθορίζουν πώς ασκούμε τα δικαιώματα επίβλεψής μας επί των προγραμμάτων. Γιατί πολλές φορές ε, έρχεται πολύ αργά η πληροφόρηση, δεν προλαβαίνουμε να την ε, αξιολογήσουμε, άρα προτείνω ένα καλύτερο σύστημα στο μέλλον για την ενημέρωση. Δεν ξέρω, Ενρίκη, αν θες να πεις κάτι σύντομα. Πότε θα μας υποβάλεις την έκθεσή σου στην Επιτροπή μας. Στο επόμενο θέμα, όπου θα μας ενημερώσει ο κύριος Γκριμό για το θέμα αυτό, θα παρέμβω και θα αναφερθώ γι' αυτό. Ναι, λέει Πρόεδρος, στο επόμενο θέμα θα έχουμε μια παρουσίαση της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης όπου θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για την ουσία των ε, θεμάτων που μας ε, ενδιαφέρουν, που είναι αρμοδιότητάς μας και όχι απλώς να σχολιάζουμε τα θέματα της ΑΦΕΤ. Όλα αυτά σχεδιάζονται με τα νέα προγράμματα και το πολιετές πλαίσιο, για τα οποία σύντομα θα μας ενημερώσει η Επιτροπή. Δεν υπάρχουν σκιώδεις για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή θέλει να μας πει τίποτα. Πολύ σύντομα παρακαλώ γι' αυτό. Συγγνώμη, ο κύριος Γκέρετς. Ναι, να κάνω μια παρατήρηση για αυτή τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτική για όλες τις προτάσεις που αφορούν την απλοποίηση της δομής του προπολογισμού. Α, Είναι το επόμενο θέμα. Το, επόμενο, το επόμενο θέμα, λέει η Πρόεδρος. Τώρα συζητάμε μόνο τη γνωμοδότηση προς την ΑΦΕΤ. Ο Μπόγκταν Βεντένα. Συμφωνούμε με την άποψή σου το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα και δυνατότητα ελέγχου. Και σας στηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Βανσάν, θέλεις να μιλήσεις τώρα για το επόμενο θέμα. Για το σχέδιο γνωμοδότησης. Τα ευρύτερα θέματα θα τα συζητήσετε στην έκθεση του κυρίου Γκερέρο για το δικαίωμα ελέγχου. Να αναφερθώ σε μερικά στοιχεία. Αναφέρεται στο σχέδιο γνωμοδότησης ορισμένα θέματα για το σεβασμό ορισμένων προθεσμιών και ελέγξαμε πώς έχει η κατάσταση και ό,τι διαπιστώσαμε πέρυσι υπήρχαν 46 εφαρμοστικά μέτρα εντός του μέσου για την συνεργασία για την ανάπτυξη που εστάλησαν στο Κοινοβούλιο για να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου με βάση τον κανονισμό για την επιτροπολογία, κυρίως ε, ετήσια προγράμματα. Από τα 46 κείμενα, μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις υπήρξε καθυστέρηση. Τέσσερις από τα 46 για την ε, αποστολή των εγγράφων. Βεβαίως οι προθεσμίες πάντα πρέπει να τηρούνται ήδη και τέσσερις καθυστερήσεις ε, είναι θέμα. Αλλά θέτει το θέμα στο σωστό πλαίσιο. Και εάν ενδιαφέρονται τα μέλη, έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόεδρος. Δεν είναι μόνο 20 μέρες είναι θέμα και πότε είναι αυτές οι 20 μέρες. Άμα μας στείλει το κείμενο αυτό στις 19 Δεκεμβρίου, δεν λέω τι συνέβη, δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι και από την Επιτροπή Ένβη, όχι μόνο εσείς, αλλά και άλλοι. Μας στέλνουν κείμενα στις 10 Ιουλίου για την ε, ενημέρωση για έναν εφαρμοστικό κανονισμό. Αυτό δεν είναι δεκτό. Υπάρχουν θέματα και αφορούν ε, πολλούς τομείς. Φιλιμπέρτο μπορεί να μιλήσει στο επόμενο θέμα. Ε, πολύ σύντομο θέμα είναι αυτό. Προθεσμία για τροπολογίες σήμερα στη μία, ψηφοφορία 25 Φεβρουαρίου, 20 Φεβρουαρίου. Ας αφήσουμε το θέμα αυτό και να περάσουμε στο πολύ πιο σημαντικό θέμα που αφορά την Επιτροπή μας. Είναι το 10 μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του μέσου συνεργασίας την ανάπτυξη και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Και να καλέσω και τον Φιλιμπέρτο να έρθει εδώ να κάτσει κοντά μας. Okay, we're running a bit behind. We have a... Ωραία, έχουμε μία σύντομη καθυστέρηση. Στις 11 και 10 θα έχουμε την κοινή συνεδρίαση με την Ίντα. Μπορεί να μας περιμένουν λίγο. Γιατί είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση το Δεκέμβριο. Υποβλήθηκαν από την Επιτροπή οι εκθέσεις για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση για όλα τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα συμπεριλαμβανομένου και του DCI και του EDF, του Ταμείου Ανάπτυξης. Οι εκθέσεις αυτές ε, υπόκειδες σε δημόσια διαβούλευση. Λοιπόν, παρακαλώ εξηγήστε τι κάνατε, πώς ε, λειτουργεί η διαδικασία αυτή και μετά θα σχολιάσουν οι συνάδελφοι. Βενσάν, μπορείς να μας εξηγήσεις εσύ. Συνάδελφοι, το Μάρτιο θα συναντηθούμε με τον Επίτροπο Νίμιτσα για τον στρατηγικό μας διάλογο όπου θα το ρωτήσουμε και τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Σήμερα όμως θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες για τα πορίσματα της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης και τι αλλαγές μπορεί να προτείνουν. Ο Βανσόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. σα παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση όσον μέσο με αξιολόγηση για αυτά τα μέσα αυτού του μηχανισμού που είναι αρμοδιότητά σα για τη συνεργασία στην ανάπτυξη, το, το DCI δηλαδή και το Ταμείο ανάπτυξη το EDF. Έχουμε ήδη κάνει σημαντική προπαρασκευή όσον αφορά το επόμενο πολιτισμικό πλαίσιο, το ώστε θα πρέπει να δούμε τώρα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία, κατάλληλοι μηχανισμοί, ούτω ώστε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία επιδέχονται βελτίωση στο μέλλον ή δυνατόν. Τώρα όσον αφορά την διαδικασία που ακολουθήσαμε για να καταλήξουμε σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτή την έκθεση ως Επιτροπή και αυτό παράλληλα συνοδεύονται κάποια έγγραφα υπηρεσιακά για την αξιολόγηση αυτών των 10 μηχανισμών που καλύπτει αυτή η έκθεση. Είναι μια μακρά διαδικασία, μας πήρε όλο το 17, είχαμε ένα σωρό διαβουλεύσεις στοχευμένες και με το Κοινοβούλιο, ανεξάρτητες αξιολογήσεις εξωτερικές που αναθέσαμε και παρουσιάστηκαν και εδώ στην Επιτροπή σας και από αυτής της βάσεως οι υπηρεσίες Επιτροπής από κοινού με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, προχώρησαν σε αυτή την προσπάθεια, αυτή τη διαδρομή. Έχουμε σε αυτό το έγγραφο και κάποια παραρτήματα για κάποια ανάλυση κατόπιν ε, έρευνας, κατόπιν ευρείας ε, διαβούλευσης, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη νομοθετική και όχι μόνο το αποτέλεσμα ότι καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Έχουν βέβαια προσωρινό χαρακτήρα, γιατί αφού μιλούμε για σαν αναπτυξιακή συνεργασία αυτή έχει μέσο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα οπότε είναι εξορισμού αυτό προσωρινό αλλά είναι και αυτό που χρειάζεται ε, για να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό πετύχαμε τους στόχους μας και να δούμε κατά πόσον έτσι μπορέσαμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια παρά το ότι θα πρέπει να δούμε επίσης αν η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε και συνέβαλε και επίσης αναδύεται από τις ερευνές μας ότι ε, έχουμε αντλήσει συμπεράσματα από το παρελθόν και έχουμε επομένω αυτά τα μέσα της συνεργασίας στην ανάπτυξη, γίνεται και διαφοροποίηση όσον αφορά την ενίσχυση, τη βοήθεια προς τους εταίρους μας. Ένα άλλο στοιχείο. Βλέπουμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί ήταν αρκετά ευρύς, ε, ευέλικτοι, οπότε θα πρέπει να δούμε ότι από την αρχή του δημοσιονομικού αυτού πλαισίου προσπαθήσαμε να έχουμε κάποια ευελιξία ούτω ώστε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Και έτσι σημειώθηκε κάποια πρόοδος όσον αφορά το mainstreaming, όσον αφορά το κλίμα και ό,τι χρειάζεται το λάβαμε υπόψη στο μέλλον και τώρα όσον αφορά τα διάφορα, διάφορα θέματα αυτής της ανησυχής συνεργασίας και προσπαθήσαμε να διδαχθούμε για το μέλλον γιατί υπάρχουν κάποιες προστριβές συγκρούσεις μεταξύ των προτεραιοτήτων ημών και των εταίρων μας και πολλές φορές αυτές οι διαφορετικές προτεραιότητες οδηγούν στο ότι η αρχιτεκτονική αυτών των προγραμμάτων είναι διαφορετική θεματικά, τοπικά ε, και αυτό προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλα αυτά που θεωρήσαμε ότι είναι ακόμα πιο κορυφαίες προτεραιότητες. επίσης έχουμε και προσθέμενη αξία από αυτήν την αντισιακή συνεργασία. Να, Φερρυπίν, σήμερα έχουμε περίπου 20% της βοήθειας που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει αυτό το 20% και φορά τη δική μας δομή για την ε, ενίσχυση. Και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτό θα αναθεωρηθεί. Και Όσον αφορά τα συμπεράσματα, θα πρέπει να δούμε τους μηχανισμούς που έχουν σχέση με τις δικές σας αρμοδιότητες, γιατί τη είναι αρμόδια και η Επιτροπή Ιστορικών Υποθέσεων. Είπαμε ότι, αυτό, ότι είναι εύστοχα αυτά τα οποία έγιναν στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου και γι' αυτό δεν προτείνεται η τροποποίηση αυτών των μηχανισμών. Υπάρχουν βέβαια περιθώρια βελτίωσης, θα πρέπει αυτά να τα λάβουμε υπόψη όταν προχωρήσουμε σε μηχανισμούς για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα τώρα στοιχείο για αυτούς τους μηχανισμούς, για την ε, χιλιετία, το είχαμε κάνει αυτό, τώρα θα πρέπει να λέμε υπόψη το θεματολόγιο 2030 και το νέο πλαίσιο μιας πολιτικής της συνένεσης γιατί θα πρέπει να προσαρμοστούν αυτοί οι μηχανισμοί στις ανάγκες του μέλλοντος στα πλαίσια του μελλοντικού πλαισίου. Είπαμε ότι έχουμε αυτή την προστριβή μεταξύ των προτεραιών ημών και των εταίρων μας. Φυσικά έχουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα εμείς ως προτεραιότητες και επίσης τις ε, αρχές και αξίες των εταίρων μας. Και άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα τι γίνεται με την κοινωνία σε εκείνες τις ε, χώρες που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ευελιξία, να καλύψουμε τα απρόβλεπτα και κάθε φορά στο πολίτες πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα και να υπάρχει περιθώριο ελιγμών διότι αλλάζει η συγκυρία. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα αποθεματικό σημαντικό όπως ε, ισχύει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη Να υπάρχει όμω και δημοσιονομικά προβλεψιμότητα και ευελιξία χρειάζεται. Άρα έτσι θα πρέπει να ζητήσουμε την ισορροπία. Προβλεψιμότητα είναι σημαντική για την ε, ενίσχυση. Προβλεψιμότητα όμως και για το πολιτές πλαίσιο και έτσι να έχουμε το απαραίτητο περιθώριο ελιγμών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνεχικότητα μεταξύ των επιμέρους μηχανισμών. Και γι' αυτό τις έχουμε ομαδοποιήσει, αναζητούμε συνέργειες και άρα προβληματιζόμαστε για το πώς θα εξορθολογήσουμε περισσότερο, πώς θα ομαδοποιήσουμε περισσότερο αυτούς τους μηχανισμούς. Είπαμε για το mainstreaming και είπαμε θα πρέπει να δούμε πώς διαρθρώνεται, πώς ταιριάζει η εσωτερική με την εξωτερική πολιτική. Πολύ σημαντικό αυτό και αυτό θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει για τους μέλλοντες μηχανισμούς. Επίσης κάτι άλλο το οποίο είναι συγκεκριμένο και αφορά την συνεργασία με τις ε, χώρες που πέρασαν από την διμερή συνεργασία και αυξήθηκε η συμμετοχή τους σε αυτή την πολιτική αλλά είπαμε δεν είναι μόνο θέμα αύξησης των πόρων. Είναι θέμα ποιοτικό. Τι συνεργασία γίνεται. Πώς θα πλαισιωθεί η συνεργασία με τις χώρες εκείνες. Α, και κάτι τελευταίο όσον αφορά τον κοινό προγραμματισμό. Εδώ θα πρέπει να θεωρηθεί θετικό ότι τώρα η φιλοδοξία μας ε, υλοποιείται να κάνουμε περισσότερα, να τα κάνουμε Α, ναι, και άλλα δύο θέματα και μια που μακρηγόρησα να σας τα πω γρήγορα, γρήγορα. Για να δούμε πώς ε, είναι η δομή τώρα του Ταμείου Ανάπτυξη. Είπαμε ότι εδώ έχουμε τη δραστηριότητα που διαρθρώνεται θεματικά και να δούμε πώς όλα αυτά θα τα συνδυάσουμε στο μέλλον. Και κάτι άλλο είναι μια ιδιορυθμία ιστορική που αφορά το EDF όσον αφορά τις περιφερειακές εθνικές ε, ε, ενισχύσεις του Ταμείου Ανάπτυξης γιατί υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που πάντοτε υπήρχε όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας προς τις εθνικές αρχές αλλά πολλές φορές ε, οι προσδοκίες δεν εκπληρώνονται. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς το μέλλον θα αναθεωρηθεί αυτό το σύστημα επί τη βάση των αρχών ε, της ικανοποίησης των αιτημάτων των ε, δικαιούχων, τόσο ώστε να πιάνει τόπο η ενίσχυση. Απ, να δώσουμε τώρα στον Φιλιμπέρτο την σκητάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ, Βενσό για αυτήν την τόσο πλήρη εισαγωγή. Οπότε να συμπληρώσω και εγώ ε, τι θα γίνει με το πολιτές πλαίσιο εν του 2020. Από πλευράς ανάλυσης μπορώ να προσθέσω ένα-δύο σημεία σε αυτά που μας είπε ήδη ο Βενσάν. Καταρχάς, αν δούμε ποια είναι η προσέγγιση πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν τη δούμε τη σκοπιά της παγκόσμιας στρατηγικής για την πολιτική περιασφαλείας βλέπουμε δύο σημαντικά στοιχεία σχετικά για τη συζήτηση. Το πρώτο είναι ότι αυτή η γενική στρατηγική δεν είναι μόνο θέμα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Είναι παγκόσμια πολιτική διότι αναγνωρίζει ότι μπορεί να πετύχει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα μόνο αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με άλλε πολιτικέ, όπω είναι η εμπορική πολιτική, η τεχνολογική πολιτική, η αναπτυξιακή πολιτική, η πολιτική συνεργασία κλπ. Ότι σταθερότητα και ασφάλεια λοιπόν της Υπήρου μας και των γειτόνων μα και των γειτόνων των γειτόνων μας εξαρτάται κατά πολύ από τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ευημερία, θέσεις απασχόλησης, ε, δυνατότητες συμμετοχής, και ε, καλή διακυβέρνηση στις χώρες εταίρους. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο λοιπόν, διότι αν θέλουμε, όπως έλεγε και ο Βενσάν, αν θέλουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον και ποια θα τα μελλοντικά μας χρηματοπιστωτικά μέσα, θα πρέπει να τα δούμε αυτά σε συνάρτηση με τη γενικότερη προσέγγιση, ούτω ώστε να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας, τις αξίες μας και θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στην παγκόσμια προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και είναι πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση για την διαμόρφωση παγκόσμιας πολιτικής. Κάτι άλλο σχετικό με τη μεσοπρόθεσμη εξολόγηση του χρηματιστοτικού μέσου είναι αυτό που ανέφερα ακροθυγός ο Βενσάν για το πόσο συνεκτικές είναι οι δράσεις μας. Στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης διαθέτουμε αρκετά μέσα. Καλύπτουμε μακροπρόθεσμες πτυχές, βραχυπρόθεσμες πτυχές, συνεργασία που συμφωνούμε με χώρες εταίρους, συνεργασία ε, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας και αυτό αυτή, ε, αυτή η πολυσχηδής προσέγγιση καλύπτει διάφορες φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αλλά ποτέ δεν τα συνδυάσαμε σωστά και τα συντονίσαμε στη σχέση που έχουμε με μια ιδιαίτερη συγκεκριμένη χώρα ή συγκεκριμένη περιοχή. Έχ... Πώς προγραμματίζουμε τα μέσα, πώς εφαρμόζουμε τα διάφορα μέσα αυτό πρέπει να εξετάσουμε. Καμιά φορά η μη σωστή χρησιμοποίησή του, μα ε, αποδυνάμωσε όσον αφορά την προσφορά που μπορούμε να δώσουμε στου τομεί που μα ενδιαφέρουν και πώ μπορούμε να πετύχουμε συμπληρωματικότητα ε, και πώ μπορούμε να προωθήσουμε σωστά τα συμφέροντά μας, αξίε μα εναντί τρίτη χώρα. Και για ένα θεσμικό όργανο όπω ε, το Ευρωκοινοβούλιο, η εποπτεία τη συνοχή και της σχέσης μεταξύ των μέσων θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. Γι' αυτό, για το μέλλον, θα εξετάσουμε τέσσερα βασικά στοιχεία. Ποιο είναι το πρώτο. Το πρώτο είναι να διαφυλάξουμε τους πόρους, το επίπεδο των πόρων για την εξωτερική δράση και κυρίως για αναπτυξιακή συνεργασία στα επίπεδα τουλάχιστον τα σημερινά και ενδεχομένω και αύξησή τους. Έχουμε πρόβλημα με τον Brexit βέβαια, οπότε θα είναι περίπλοκο θέμα η κατάρτιση του προπολογισμού και το ανώτατο όριο, αλλά η διαφύλαξη του σημερινού επίπεδου, η αύξηση του σημερινού επίπεδου βοηθείας που παρέχουμε σε τρίτες χώρες είναι σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη το 0,7% που είναι στόχος κοινό μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και πιθανότατα και τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν, όχι μόνο το Κοινοβούλιο, την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης και σημασία να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο χρηματοδότηση. Αυτό το πρώτο. Δεύτερον, συνοχή και απλούστευση. Κάτι που συνδέεται με τα προαναφερθέντα. Πιστεύουμε ότι θα είχε αξία να μειώσουμε τον αριθμό των μέσων, να τα συνδυάσουμε και τα συμπτύξουμε στο βαθμό του δυνατού, ούτω ώστε να τονίσουμε όλος ιδιαίτερο την κοινή προσπάθεια Χρήση των διαφόρων πολιτικών και των προσφορών μας περί συνεργασίας με άλλες χώρες. Ε, ένα ευρύ πεδίο μέσων και διαφοροποιημένα μέσα είναι κάτι που απαιτεί διαχείριση. Πρέπει να προβλέπουμε το πώς θα γίνεται η κατανομή για διάφορες περιοχές και διάφορες ομάδες, να προστατεύουμε τα συμφέροντά μας βέβαια, σχέση με τους εταίρους, λεπτομέρειες εφαρμογής προγραμμάτων μακροχρόνιος προγραμματισμός, ίσως χρειάζεται όμως και βραχυπρόθεσμη άμεση δράση, λεπτομέρειες διαμόρφωσης εφαρμογής που επιτρέπουν ταχεία προσαρμογή. Ίσως για εφαρμογή ε, ίδιας πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να μπορούμε να κινούμεθα πιο γρήγορα σε συνεργασία με άλλες χώρες. Ταυτόχρονα λοιπόν μπορούμε να συνδυάσουμε τεφιστάμενα μέσα και να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τη δυνατότητα που έχουμε να καθησυχάζουμε και να εγγυόμεθα ε, στους εταίρους μας τι προσδοκίες μπορούμε να έχουν απέναντί μας και να διαφυλάσσουμε τα συμφέροντά μας και να προωθούμε και τις αξίες μας. Μετά άλλο σημείο, η ευελιξία. Στις παρούσες δημοσιονομικές προπτικές αυξήσαμε στο μέγιστο δυνατό το αποθεματικό και την ευελιξία του, ε, του προϋπολογισμού στην τελευταία μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των δημοσιονομικών προπτικών είχαμε σημαντική μετακίνηση πόρων προς την εξωτερική δράση, 3,9 ε, δις περισσότερα, αλλά αυτά τα στοιχεία της ευελιξίας δεν αρκούν. Και το παράδειγμα που δόθηκε για την ένταξη στον προπολογισμό της ευελιξίας που υπάρχει στο ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και να υπάρχει και σημαντικό απόθεμα ο πολιτής χαρακτήρας των πιστώσεων και πώς ήδη να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αναλήψεις υποχρεώσεων, να τις αναδιατάξουμε, ε, είναι πολύ σημαντικά για μελλοντικά χρηματοπιστωτικά μέσα. Τέλος. το πώς υποβάλλονται οι εκθέσεις οι διάφορες, πώς μπορούν να ελέγχονται και να καταλογίζονται οι πιστώσεις. Αν δούμε την ευελιξία της εξωτερικής δράσης, έχουμε 96% των πόρων όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Λοιπόν, να δούμε πιστασισμένος μέσος όρος μεταξύ των απαιτήσεων που υπάρχει κάθε μέσο. Υπάρχει διαφοροποίηση για τα διάφορα στοιχεία διάφορα στοιχεία, διάφορα μέσα. Έχουμε διαφορετικό επίπεδο ε, υποβολής απαιτήσει για εκθέσεις για την αντιξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να εντοπίσουμε στο μέλλον λοιπόν τη σωστή αρχιτεκτονική που απαιτείται. Ίσως ένα επίπεδο ε, ενημέρωσης που θα πρέπει να πετύχουμε και ό,τι γίνει παραπάνω από αυτό θα είναι βελτίωση. Είμαστε στο 96% παρόλο που δεν έχουμε δεν ε, έχουμε αυτή τη νομική υποχρέωση. Δεν τίθεται σαν νομική υποχρέωση. Τώρα ένα σχόλιο στην πρώτερη συζήτηση. Ε, από την πρόσφατη εμπειρία που είχα τα τελευταία δύο χρόνια μπορώ να πω ότι στον το στρατηγικό διάλογο και την προετοιμασία του στρατηγικού διαλόγου μέσω εγγράφων και στα πλαίσια των κανόνων ε, στα πλαίσια τα χρονικά για να μπορείτε να διεξαγάγετε τον έλεγχό σας, τα πράγματα πήγαν ικανοποιητικά. Τι θέλω να πω, ότι είμαστε στη διάθεσή σας. για το διάλογο αυτό να διευκολύνουμε τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και να τον ε, βελτιώσουμε, να γίνει καλύτερος από ό,τι είναι σήμερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Για το συνάδελφους της ΣΥΝΤΕ, κοιτάξτε, μείναμε λίγο πίσω Μιλάμε για σημαντικά θέματα που μπορεί να είναι ενδιαφέροντα. Μιλάμε για, το, για τη μελλοντική μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, για τα μελλοντικά μέσα, τα μεγάλα μέσα που καλύπτουν τι εξωτερικές δράσεις και είναι θέματα που ενδιαφέρουν δεχομένω και τους ε, συναδέλφους για τα, που εξετάζουν τα εμπορικά ζητήματα. Ζητάν συνάδελφοι το λόγο. Ο Φρανκ Έγγελ έχει πρώτος το λόγο. Merci, Linda. Ευχαριστώ Λίντα. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις που ακούσαμε από τον αμιλητή. Το θέμα είναι, είναι πάντα σημαντικό, φορά την κατάρτιση, το σχεδιασμό του προπολογισμού και για αυτούς που είναι αποδέκτες ε, είναι στοιχεία που τους έλειψαν. Άλλη φορά που τους ήρθα σε επαφή μαζί τους μου είπαν αν μπορείτε να μας πείτε αν έχετε πραγματικά την πρόθεση κάθε μήνα να μας χτυπάτε, να μας πλήττετε με ένα νέο μέσο και πρέπει να μαθαίνουμε πώς λειτουργεί. Όπως ήταν τότε το Ταμείο για Εξωτερικές Επενδύσεις που ήταν το νέο μέσο που είχε δημιουργηθεί. Θεωρώ ότι είναι κατανοητό ότι έχουμε την παρούσα κατάσταση να αντιμετωπίσουμε, διότι θεωρώ ότι τη στιγμή που ξεκίνησε η περίοδος του οικονομικού σχεδιασμού, στον οποίο βρισκόμαστε, κανείς δεν ονειρεύτηκε μια τόσο μεγάλη μεταναστευτική κρίση και το μεταστατικό φαινόμενο με όλες τις πτυχές αυτού μας οδήγησε να εφευρίσκουμε καθοδόν κάποια πράγματα ε, για τα οποία δεν υπήρχε συγκεκριμένο μέσο ούτε πραγματικά επαρκής χρηματοδότηση. Και προσπαθούμε λοιπόν ε, ε, ε, να παίζουμε με τα στοιχεία και με τα εκατομμύρια, να δώσουμε την εντύπωση ότι χρηματοδοτούμε κάποια διαδικασία στην Αφρική που θέλουμε επιτόπου να την ενισχύσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ενισχύουμε τίποτα. Ένα από τα στοιχεία που παρουσιάζονται, ξέρω, είναι αξιόπιστα. Λοιπόν, από αυτά παρουσιάζονται, τα στοιχεία μας λένε ότι για να επιτρέψουμε στην Αφρική ανάπτυξη υποδομών σε λογικό επίπεδο χρειαζόνται 70 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ε, έτη φωτός απέχουμε εμείς ε, και κυρίως σε συγκρίση με τους Κινέζους, τους φίλους μας. Εγώ δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, ε, να μιμηθεί άλλες προσεγγίσεις αλλά περισσότερη ταχύτητα σε αυτή τη διαδικασία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα χρειάζεται, χρειάζεται αξιοπιστία. Θα ήταν καλό κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρο ότι μέσα στα θέσιμα μέσα στη διάσκεψη των δωρητών στην Κεντρική Αφρική 2,3 δισεκατομμύρια είχαμε υποσχεθεί. 10% έχουμε δώσει από αυτά μέχρι τώρα στην πραγματικότητα. Πώς θέλουμε εμείς να μας πάρουν στα σοβαρά οι συνομιλητές όπως εκεί που είναι οι πιο φτωχοί των φτωχών, που δεν έχουν φίλους παρά μόνο μας. Αν υποσχόμεθα ε, κάτι που δεν τηρούμε. Και δεν θα ήταν κάτι που θα έκανε το προπολογισμό μας να καταρρεύσει, αν τηρούσαμε τις υποσχέσεις μας. Τελευταία λοιπόν ε, σκέψη που ανήκει στον τομέα συνοχής και αξιοπιστίας, ιχνηλασιμότητας, δεν ξέρω πώς θα το πούμε αλλά και αξιοπρεπίας. Ανοίξει την πτυχή της αξιοπρέπειας. Θα πρέπει να δούμε ε, τι κάνουμε λοιπόν όσον αφορά ε, τις υποχρεώσεις που έχουμε. Αν θέλουμε αυτή η συνεργασία, κυρίως με την Αφρική, και αφορά τι γίνεται μετά το Κοτονού, μετά το 2020 σχέσεις. Αν θέλουμε να γίνει στρατηγικός εταίρος η Αφρική, κάτι που επαναλαμβάνουμε συνεχώς όταν μιλάμε, θα πρέπει, πιστεύω, αυτή η συνεργασία να δράζεται περισσότερο επί αξιοπιστίας, αξιοπιστίας των παροχών μας, των επενδύσεών μας, αν θέλετε, στην Αφρική, αλλά και επί της ε, ελευθερίας που θα έχουν οι χώρες Αφρικής, πώς θα διαθέτουν αυτούς τους σπόρους στα πλαίσια λοιπόν της λογικής ε, της ε, μελλοντική προσέγγισης που ακολουθήσει η Αφρική για την εξέλιξή της. Νομίζω, ξέρουμε τι δεν είναι ιδεώδες μέχρι τώρα, ότι χρειάζονται ακόμα περισσότεροι, περισσότεροι πόροι στους μελλοντικούς ε, σχεδιασμούς. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου, αλλά δεν ξέρουμε τι θέση θα έχουν τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά αυτά τα στοιχεία αποτελούν συνιστώσεις μιας πιο ορατής, πιο λογικής, πιο ενισχυτικής αν θέλετε πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως που μας οδηγεί προς το στόχο ε, που είναι μια ε, περισσότερο πολιτική συνεργασία παρόχι και όχι πολιτική συνεχούς εξάρτηση. Ο κ. Γκερέρο που θα είναι συγκητής μας για την έκθεση εφαρμογή των ε, προγραμμάτων θα πρέπει να πάρει το λόγο. Bueno, gracias. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα έχουμε την πρώτη μας προσέγγιση των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ και τον κύριο Έγγελ για τα όσα μας είπε. Σήμερα ήρθε εδώ ο κύριος Φιλμπρίτε και ο κύριος Γκριμό και ακριβώς γιατί βρισκόμαστε στην διαδρομή της σύνταξης αυτής της έκθεσης που θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Όπως σας είπα, πρόκειται για εφαρμοστική έκθεση. Αυτό πάει να πει ότι περιέχει και κάποια αξιολόγηση για το πώς λειτουργήσαν οι μηχανισμοί μέχρι σήμερα, πώς εφαρμόστηκαν. Ταυτόχρονα όμως όλα αυτά αυτά γίνονται σε μια συγκυρία οπότε προετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Μάιο. Τότε θα παρουσιάσει την πρόταση για ε, την επόμενη ε, το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιετές όσον αφορά τους πόρους της Ένωσης, όσον αφορά τους μηχανισμούς με τους οποίους η Ένωση πρόκειται να υλοποιήσει τις πολιτικές της. Ε, γι' αυτό η έκθεση αυτή γίνεται από τη μια μεριά μια έκθεση αξιολόγησης αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί και μια αξιολόγηση της Επιτροπής μας για το πώς θέλουμε να βλέπουμε την Επιτροπή σύμφωνα με την πολιτική ανάπτυξη και τι γίνεται με τους μηχανισμούς υλοποίηση αυτής της πολιτικής στα πλαίσια του πολιετούς πλαισίου όπως είπε και η Πρόεδρος. Έχουμε ταυτόχρονα και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που συντάσσει άλλη έκθεση όσον αφορά τους γενικούς μηχανισμούς της εξωτερικής ε, πολιτικής. Και ήρθα σε επαφή με την Μαριέτε Σάχτα και προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα συντονιστούμε. Πώς δηλαδή θα συνδυαστεί η διαδρομή αυτών των δύο εκθέσεων. Ακόμα δεν έχω διαβάσει την έκθεση εκείνη, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μπορέσουμε να τους πούμε τη δική μας βασική θέση το ότι δηλαδή θέλουμε να περιφρουρηθεί η ταυτότητα, οι αξίες και οι μηχανισμοί της πολιτικής ανάπτυξης στα πλαίσια αυτής της ε, εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κάποια στιγμή όταν μας μίλησε ο κύριος Φιλιμπέρτο το είπε. Μας είπε μέχρι ποιο σημείο η πολιτική ανάπτυξη είναι σημαντική για την εξωτερική στρατηγική της ε, Ένωσης. Μια αν αυτό το οποίο θέλουμε να είναι να εξασφαλίσουμε σταθερότητα και ασφάλεια ε, γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αυτό κατά πολύ θα επιτευχθεί από αυτό που ονομάζουμε soft power, δηλαδή τη δυνατότητα της Ένωσης να μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη, στην διακυβέρνηση, να προλαβαίνουμε τις ε, συγκρούσεις και τις προστριβές, να επιλύουμε τις συγκρούσεις που ξεσπούν γύρω μας. Επίσης, είχαμε και κάποιες επίσημες συναντήσεις με τον Επίτροπο Νίμιτσα, οπότε και θα πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Γκριμό. Ε, χτες είχαμε αυτή την συνάντηση και έγινε έτσι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το πώς απέδωσαν μέχρι σήμερα αυτοί οι μηχανισμοί, αυτοί που αναφέραμε. Είπα εγώ το ότι ναι λειτουργήσαν αποδοτικά, ικανοποιητικά, όμως θα πρέπει να προσαρμοστούν αυτοί οι μηχανισμοί στις αλλαγές της παγκόσμιας ε, συγκυρίας. Μα έχουμε αλλαγές όμως και στη δική μας πολιτική ανάπτυξη όσον αφορά τους βιώσιμους στόχους ανθρωπιστικά, όσον αφορά το κλίμα κλπ. Άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ευελιξία αλλά και την προβλεψιμότητα και βιωσιμότητα και να κάνουμε περισσότερα στον κοινό προγραμματισμό. Να προσαρμόσουμε τις προτεραιότητές μας στα όσα απαιτούνται, στα όσα ζητούνται από τους εταίρους μας. Γι' αυτό έχω να σας πω το εξής. Η έκθεση την οποία θα σας προσφέρω στην επόμενη συνάντησή μας ε, θα έχουμε τρεις άξονες. Ε, στην παρουσίαση αυτή πρώτα πρώτα αξιολόγηση αυτών των μηχανισμών. Το δεύτερο άξονα θα συζητήσουμε για το τι προσδοκούμε από την ε, εφαρμογή αυτών των μηχανισμών στο υπόλοιπο που μένει που ισχύουν αυτοί οι μηχανισμοί και τρίτον να δούμε για το πώς θα θέλαμε η Επιτροπή μας να πλαισιωθεί από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρόταση για την επόμενη περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών. Και τώρα θέλω να επανέλθω στα όσα μας είπε ο κύριος Φιλιμπέρτο. Ε, βέβαια και θέλουμε εμείς να παραμείνουν ή και να αυξηθεί η πρικοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, και έτσι να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του Brexit να συμβάλλει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη. Εντάξει, δεν είμαστε αντίθετοι στον υπάρχει κάποια πλούστευση των μηχανισμών. Τα είπε και ο κύριος Γκέρενς. Όχι, όχι, δεν είμαστε κατά της απλούστευσης. Όμως, η ιδιωτυπία της ε, πολιτικής ανάπτυξης θα πρέπει να αναδεικνύεται κάθε φορά που έχουμε κάποιον νέο μηχανισμό. Ε, βέβαια και όλα αυτά εντάσσονται στην εξωτερική πολιτική Ένωσης, αλλά δεν θα πρέπει να υποταχθούμε κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την πολιτική. Θα πρέπει ε, να λαμβάνεται υπόψη αυτή η ιδιοτυπία, η ιδιορυθμία, η μοναδικότητα της Επιτροπής Ανάπτυξης, όπως τα είπε και ο κύριος Έγγελ. Χρειάζεται ευελιξία και έτσι να μπορούμε να ενεργήσουμε εν ώψη κάποιων απροβλέπτων. Όμως, πέραν των θεσμικών οργάνων, έχουμε την κοινωνία, έχουμε τις ΜΚΟ, όλοι αυτοί είναι εμπλεκόμενοι στην, ε, ε, στην πολιτική της αναπτυξής, οπότε θα πρέπει όλοι αυτοί να μπορούν να εντάσσονται ε, μέσω του προγραμματισμού μας στην αναπτυξιακή δράση. Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε στο τι γίνεται με τους ε, πόρους για την ανάπτυξη και πέραν των εισηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δούμε το πώς θα αναδειχθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου, ο ρόλος της επιτήρησης, της εποπτείας. Όλα αυτά τα πούμε στην έκθεση. Να μην επεκταθώ κι άλλο θα μπορούσα, όμως θα πρέπει τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερο χρόνο στις επόμενες συναντήσεις μας. Ε, γιατί τώρα υπάρχει πίεση μια που έχουμε αυτή την κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Σας είπα μόνο βασικά, τα πιο σημαντικά Καλά, καλά, καλά. και πρόκειται να επανέλθουμε στο θέμα τη δική σου έκθεση και τότε θα μα διατυπώσετε τι προτάσει σου για το μέλλον. Ποιο άλλο ε, θέλει το λόγο. Α, θέλετε να δευτερολογήσετε, κύριε Γκέραντ. Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι τώρα περιμένουν οι συνάδελφοι τη ε, ΙΝΤΑ. Και εξάλλου θα επανέλθουμε στην έκθεση, κύριε Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Και είμαστε, είμαστε περίεργο θεσμικό όργανο. Αποφασίσαμε ως Επιτροπή να στηρίξουμε αποφασιστικά την Κομισιόν που θέλει να εισαγάγει τις αρχές διαφοροποίησης. Να δίδονται οι χρηματοδοτήσεις στις χώρες που τις έχουν τη μεγαλύτερη, τη μεγαλύτερη ανάγκη και όχι σε χώρες που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και τι διαπιστώνουμε τώρα? Το αντίθετο. Θα δώσουμε λεφτά στην Τουρκία προς, σε χώρες που δεν είναι πλέον αναπτυσσόμενες, που θα περάσουν σε μέσο επίπεδο ανάπτυξης. Αλλάζουν λοιπόν οι προτεραιότητές μας και πηγαίνουν ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση της αρχής της διαφοροποίησης. Και το κάνουμε, συνηθίζουμε να το κάνουμε και εκπλήσουμε που δεν προκαλεί καμία συζήτηση. Πρέπει να ξαναδούμε την κατάσταση, να ξαναδούμε τις αρχές τη διαφοροποίησης. Ή θα συνεχιστεί η τρέχουσα κατάσταση που αλλάζει την ε, προηγούμενη και είναι αντίθετη με αυτά που έχουμε ψηφίσει. Και κάτι άλλο για να τελειώνω, Πρόεδρε. Εγκρίνουμε προπολογισμού. Αν θα έπρεπε να δώσουμε Όσκαρ για τον παραλογισμό, τότε θα έπρεπε να το λάβει η διαδικασία έγκρισης ε, του προπολογισμού της Ένωσης. Κάθε τρει μήνες, λέμε, δημιουργούμε ένα νέο καταπίστευμα. Υπάρχει πληθώρα χρηματοδοτικών οργάνων που ελέγχονται κατά το μάλλον και ήτον από το Κοινοβούλιο και επίσης η Επιτροπή παζαρεύει με τα κράτη-μέλη για να βοηθήσουν με ποσά που δεν θέλουν να δώσουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και όπως είπε ο κ. Σέγγελ, στα τελευταία ανάλυση δεν δίνουμε αρκετά. Το χάσμα μεταξύ των υποσχέσεων χρηματοδότησης και της πραγματικής χρηματοδότησης ε, είναι βάραθρο. Αυτό μειώνει την αξιοπιστία μας. Να κάνουμε μια πιο αποφασιστική πρόταση για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και να πούμε όλες οι χρηματοδοτήσεις θα περνάνε από τον ενωσιακό προϋπολογισμό και αν χρειάζεται κάποιο επιχείρημα για να αυξηθεί ο προπολογισμό, αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτό που μόλι εξήγησα. Ξέρω δύο χώρε που είναι διατεθειμένες να πληρώσουν περισσότερα στον προπολογισμό. Η Ουγγαρία και η Πολωνία. Ε, Α τι υποχρεώσουμε να τηρήσουν τι υποσχέσει του και να πείσουμε και τι άλλε. Γιατί όπω πάνε τα πράγματα τώρα, είναι η αρχή του τέλους μιας ε, μακράς διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μια πολιτική ανάπτυξη καινή περιεχο, περιεχομένου. Και ξέρετε ότι με τον ε, συνηθισμένο ανεδίμου τρόπο είπα ότι αυτά που υπόθηκαν για την βούληση των... αυτά που είχα πει εγώ τότε για το κατά πόσο υπάρχει βούληση τήρησης των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων ισχύει ακόμη. Πρέπει όντως να πείσουμε τα κράτη-μέλη να τηρούν τις υποσχέσεις που διατυπώνουν επισήμως σε συμπεράσματα του Συμβουλίου, σε επίσημες ομιλίες της Ένωσης από πλευράς των κρατών μελών στην Αντίσα Μπέμπα και αλλού. Ανησυχώ ιδιαίτερα για τις τελευταίες εξελίξεις στην κατεύθυνση της πολιτικής ανάπτυξης. Πρόεδρος, ε, συνάδελφοι, θα επανέλθουμε πολύ πιο αναλυτικά για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι η Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, κατάλαβαν τις ανησυχίες μας. Πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα για την πολιτική ανάπτυξης είναι μακροπρόθεσμη. Και τα καταπιστεύματα βεβαίως ε, τελικά εξυπηρετούν την ανάγκη ευελιξίας την ανάγκη δηλαδή να αντιδράσουμε σύντομα σε νέες καταστάσεις. Σας παρακαλώ να απαντήσετε σύντομα. Ένα λεπτό ο καθένας γιατί περιμένουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το θέμα της μεταναστευτικής κρίσης και την ευελιξία που μας επέτρεψε να την αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς επειδή υπήρξε ευελιξία στον, ε, στο Ταμείο για την Ανάπτυξη, καταφέραμε να καταλήξουμε περίπλοκες ε, διαπραγματεύσεις με τη Συρία και την ε, Τουρκία. Αν δεν υπήρχε αυτή η ευελιξία θα είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες όπως ισχύουν. Δεύτερον, για μεγάλο χρονικό διάστημα Η Ένωση ε, δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τα καταπιστεύματα όπως τα αξιοποιούσαν άλλοι. Μόνο με, στην την εργαλειοθήκη ε, το 12-13 ε, μπορούμε να το κάνουμε. Και έκτοτε έχουν δημιουργηθεί τέσσερα καταπιστεύματα, όχι ένα κάθε τρεις μήνες. Εντάξει, μπορεί να έχει κανείς άποψη συγκεκριμένη για αυτά τα μέσα, αλλά δεν είναι δυνατόν να πει κανεί ότι υπάρχει πληθώρα καταπιστευματών. Είναι ανακριβέ. Κάτι άλλο για την διαφοροποίηση και το 0,7% διαφοροποίηση. Να δούμε τα στοιχεία. Η Τουρκία πάντα ήταν ε, η πρώτη δικαιούχο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμη. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Τώρα για τη συγκέντρωση πόρων για τι πιο ευαίσθητε χώρε. Είναι θέμα ακριβώ αυτό κάνουμε. Αν δούμε τα στοιχεία θα δείτε ποιε χώρε χρηματοδοτούμε. Και για το 0,7% βεβαίω συμφωνώ. Τα κράτη-μέλη τη Ένωση επανέλαβαν αυτή τη δέσμευση. Όταν θα υπάρξει συζήτηση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να τηρηθεί αυτή η υπόσχεση. Φιλιμπέρτο, έχει να προσθέσει τίποτα άλλο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο βουλευτή που είπε ότι η αναπτυξική πολιτική δεν θα πρέπει να είναι απλώς τμήμα της ε, εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι η παγκόσμια στρατηγική που προωθούμε ακριβώς αυτό σέβεται. Θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να βοηθήσουμε τους ε, εταίρους μας να γίνουν βιώσιμοι. Αυτό είναι βασικό στοιχείο της εξωτερικής μας ε, πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να συμβαδίζουν τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντα των εταίρων μας όχι το ένα να υπερισχύει του άλλου. Για την έλλειψη πόρων και την ε, από αυτούς ε, θεωρούμενη έλλειψη αποτελεσμάτων. Όχι, δεν υπάρχει πληθώρα νέων μέσων. Απλώς χρησιμοποιούμε περισσότερο αυτό το συνδυασμό, αυτό το blending ε, μέσω επενδύσεων από ιδιωτικού φορείς, μέσω περισσότερης χρήσης ε, εγγυήσεων ή την ε, ε, συνδυασμένη τεχνική και χρηματοδοτική και βοήθεια σε επίπεδο πολιτικής. Αυτός είναι ίσως ο πιο σημαντικός τρόπος για να καλυφθεί αυτό το κενό μεταξύ των διαθέσιμων και των αναγκαίων πόρων. Νομίζω ότι το blending μέχρι στιγμής τα έχει πάει καλά. Δεν ξέρω απ' έξω τα στοιχεία αλλά με μερικές δεκάδες ε, εκατομμυρίων μέσω του blending, μέσω του συνδυασμού και με ιδιωτική χρηματοδότηση, είχαμε μία μόχλευση επί 10, επί 12. Επενδύθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Ελπιδοφόρος λοιπόν ε, προοπτική. Είμαι κάπως ε, λιγότερο απεσιόδοξος. το πώς αξιολογώ τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει. Νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών έχει ως αποτέλεσμα ότι είμαστε ο πρώτος χορηγός παγκόσμια αναπτυξιακής βοήθειας. Ναι, μεν δεν τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας το 2015 από πλευράς δεσμέσων, αλλά αυξάνεται η συλλογική μας επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και υπάρχει αυτή η δέσμευση, όπως υπόθηκε, για το 0,7 πρόοδος Ευχαριστώ πολύ. Σαλ, όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται. Η συνάδελφοι τη ΙΝΤΑ. Όχι, όχι, όχι. Μα δεν κατηγόρησα κυρίω τα καταπιστεύματα, τα οποία στήριξα ζήτηση. Αυτό που επικρίνω είναι η απίστευτη και ανεύθυνη στάση των κρατών μελών που κάνουν δηλώσεις, δεν, δεν τηρούν τις υποχρέσεις τους, αντί να κάνουν δηλώσεις να αυξηθεί ο ευρωπαϊκός προπολογισμό και όχι η Κομισιόν να πηγαίνει να παρακαλάει να εκετεύει τα κράτη-μέλη. Ε, το θέμα αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να, υπάρξουν, να υπάρξει το νέο πολιτέ πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα. Είμαι σίγουρο ότι θα επανέλθετε όταν θα παρουσιάσει την έκθεσή του ο κύριο Γκερέρο. Θα είστε καλοδεχούμενοι. Συγγνώμη για του συναδέλφου τη ΙΝΤΑ ε, που καθυστερήσαμε. Θα καλέσω τον συμπροεδρό μου να συμπροεδρεύσει.